Good afternoon, dear colleagues, dear guests. We will start our... συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τις συνεδρίες της Επιτροπής μας. Και θα συνεχίσω στα λιθουανικά. Παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κρίνουμε την ημέρησα διάταξη. Το σημείο 5 στην ημέρησα διάταξη για με την ανταλλαγή απόψεων με την υπερασπίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Κουρδιστάν. Ε, ε, έχει τροποποιηθεί ε, δυστυχώς το βίντεο μήνυμα που θα μας έστελνε είναι, δεν μπορούσε να έρθει ε, θα την ε, αργαστήσει Σιρπίλ και Μάλμπι που θα αντικαταστήσει λοιπόν τη Λέιλα ε, η οποία δυστυχώς είναι ασθενής εάν δεν υπάρχουν σχόλια να συνεχίσουμε τις εργασίες. Εγκρίνεται με στη διάταξη προφανώς. είναι παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα μονάχα να ξεκαθαρίσω ότι η Λέιλα Κουβάνο προφανώς δεν μπορεί να είναι παρούσα γιατί ε, βρίσκεται σε πάρα πολύ κακή θέση ε, λόγω της απεργίας πείνας την οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς, εδώ και πολλούς μήνες. Ε, αυτό ήθελα να σας πω. Ačiū. Ačiū tikrai už informaciją, linkim jai Ευχαριστούμε για αυτή την πληροφορία. Σε ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης της 20 Φεβρουαρίου, 27 Απριλίου μια σειρά από συνεδριάσεις σε του 2018 καθώς 23 Ιανουαρίου 2019 Φεβρουαρίου 2019, καθώς και 7 Μαρτίου 2019. Νομίζω ότι μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά αυτά. Και περνάμε τώρα στο σημείο 3, ανακοινώσει του Προέδρου. Στη συνεδρία είμαστε 27 Φεβρουαρίου. Οι συντονιστές αποφάσισαν στα πλαίσια της δημοσιονομικής διαδικασίας για το 2020 να δώσουν στην ομάδα του ΕΛΚ την έκθεση. Επίσης θέλαμε να καλωσορίσουμε μια ομάδα επισκεπτών της Ευρωβουλευτού της κυρίας Νόιχελ από μια οργάνωση γυναικών της, από το SPD από τη Γερμανία. Σημείο 4 τώρα. Ο ρόλος των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες. Σήμερα προβλέπεται μία ακρόαση συμμετοχή των γυναικών στην πρόληψη σειράξεων και στην επίλυση ε, ένοπλων σειράξεων, οι γυναίκες μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά ε, στην επίλυση τέτοιου είδους διαφορών και βεβαίως υπάρχουν και επιπτώσεις μιας ένοπλης σύραξης. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το ρόλο των γυναικών και την ανάγκη συμμετοχής τους και στο πώς μπορούν να συνεισφέρουν θα αφιερώσουμε ένα μέρος της ακρόασης αυτής ε, στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Έχουμε καλέσει εδώ πέντε εμπειρογνώμονες. Θα ακούσουμε, θα δούμε και την παρουσίαση μιας μελέτης που ζητήθηκε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα θα δώσω το λόγο στην Γιώχανα Πότανεν που είναι επικεφαλής ε, της των γυναικών ειρηνευτριών. Ε, είναι πραγματικά χαρά και τιμή μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ επίσης ε, που οργανώσετε αυτή την ακρόαση για αφορά ένα ζήτημα εξαιρετικά επίκαιρο. Να πω δύο λόγια για, τον εαυτό μου αλλά και για την οργάνωσή μου. Προέρχομαι από την πρωτοβουλία διαχείρισης κρίσεων που είναι μια ανεξάρτητη φιλανδική οργάνωση ε, που προσπαθεί να επιλύσει αλλά και να προλάβει ένοπλε ε, βίες σειράξει μέσω του διαλόγου και τη διαμεσολάβηση. Το 2000 οργανώθηκε, δημιουργήθηκε αυτή η οργάνωση από τον, τον πρώην πρόεδρο τη Φιλανδία, τον Μάρτι Αχτισάρη ε, και έχουμε εργαστεί σε 10 ειρηνευτικέ διαδικασίε κυρίω στην Ευρασία, στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά του CMI, λοιπόν, τη οργάνωση αυτή, η ενίσχυση και η υποστήριξη του ρόλου των γυναικών σε αυτές τις διαδικασίες είναι προτεραιότητα. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις αξίες μας, έχει να κάνει και με το ότι πραγματικά πιστεύουμε ότι αυτός είναι ένας τρόπος να ενισχυθεί ε, η προσπάθεια που κάνουμε για την επίλυση ε, των ε, βίων συγκρούσεων. Το κάνουμε αυτό με δύο τρόπους. Ενισχύουμε τις δυνατότητες διαμεσολάβησης για ζητήματα που φορούν τα δύο φύλλα, των ανθρώπων, των οργανώσεων που προετοιμάζουν αυτές τις ειρηνευτικέ διαδικασίες. Επίσης, δίνουμε εστιασμένη ενίσχυση σε γυναίκες που έχουν πληγεί από αυτές τις σειράξει. Ε, έτσι λοιπόν, σε μεγάλο βαθμό βασίζεται αυτό που θα πω στις εργασίες μας, στις υπάρχουσες ε, εξελίξει ειρηνευτικέ διαδικασίε. Γιατί λοιπόν έχει τόσο μεγάλη σημασία το θέμα αυτό. γιατί είναι σημαντικό να συμπεριλαμβάνονται οι γυναίκες σε αυτή τη διαδικασία επίλυσης διαφορών. Ε, υπάρχει βεβαίως το ψήφισμα του ΟΗΕ, ε, υπάρχουν και άλλες ακόμα, άλλα ακόμα επτά ψηφίσματα και διεθνές ε, δεσμεύσεις όπως το ΣΥΜΠΑ, όπου ε, δηλαδή σε ρυθμιστικό, σε θεσμικό επίπεδο είναι κάτι το οποίο έχει ήδη τονιστεί. Αυτό είναι μία πτυχή μόνο. Όμως το θέμα είναι ποιος είναι αυτός ο οποίος οικειοποιείται την ειρήνη την οποία θέλουμε να πετύχουμε. Ε, ποιος αναλαμβάνει τη δέσμευση σε εθνικό επίπεδο. Ε, είναι θεμητή αυτή η προσπάθεια στα, μάτια όλων των πολιτών ή μόνο για αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στην ενόπλη σύραξη. Ε, λαμβάνει η χώρα και μια κάποια έρευνα, εμπειρική έρευνα, για το πώς θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν οι γυναίκες στις συζητήσεις ε, και πώς αυτή η συμπερίληψη διευρύνει το πεδίο της συζήτησης, δίνει νέες προοπτικές, αναφέρεται ε, σε άλλες ανάγκες, σε ε, άλλες ε, προσεγγίσεις. Αυτός είναι ένας λόγος ε, για μεγαλύτερη συμπερίληψη, μεγαλύτερη συμμετοχή, να ξέρουμε τελικά τα συμφέροντα και οι ανάγκες ποιων ε, εξυπηρετώνται με αυτές τις διαδικασίες, διότι αφήνοντας απ' έξω τον μισό πληθυσμό λείπουν δράστε, λείπουν παράγοντε οι οποίοι μπορούν πραγματικά να συνεισφέρουν σε την ειρηνευτική προσπάθεια. Το βλέπουμε ε, στην Ιεμένη, παραδείγματο χάρη. Συχνά οι γυναίκε είναι αυτέ οι οποίε έχουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, έχουν γίνει και ανταλλαγέ ε, κρατουμένων ε, λόγω που το έχουν οργανώσει οι γυναίκε επειδή έχουν καλύτερη πρόσβαση. Εάν δεν το λάβουμε υπόψη μα και το προσέξουμε αυτό, είναι σαν να μην κάνουμε καλά τη δουλειά μα. Βεβαίω υπάρχει και ένα πιο μακροπρόθεσμο ζήτημα ειρηνευτικέ διαδικασίε αφορούν κάποιε στιγμές στην ιστορία όπου ε, μπορεί να κανείς να ξαναγράψει ουσιαστικά τους κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού. Και όταν ε, αυτοί οι κανόνες γράφονται με βάση και την ισότητα των δύο φύλων, τότε θα είναι και πιο μακροπρόθεσμες και πιο ε, βιώσιμες. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό για, μια, για πιο δημοκρατικέ κοινωνίε, κοινωνίε κοινωνίες που λαμβάνουν περισσότερο την ισότητα των δύο, υπόψη την ισότητα των δύο φύλων. Ε, υπάρχουν μακροπρόθεσμοι λόγοι λοιπόν, αλλά και πολλοί βραχυπρόθεσμοι, πρακτικοί λόγοι για τη συμμετοχή των γυναικών σε αυτέ τι διαδικασίες. Στην πραγματικότητα όμω, ε, έχουν περάσει 20 χρόνια από το ψήφισμα εκείνο, το πρωτοπόρο, και αν δούμε τι ερευνητικέ διαδικασίε ανά τον κόσμο, δεν βλέπουμε μεγάλο αντίκτυπο το ψήφισμα 13-25 θεωρείται ε, ότι είναι από αυτά τα ψηφίσματα για τα οποία έχουν υποθεί πολλά, αλλά έχουν γίνει πολύ λίγα. Έχουν γίνει κάποια πράγματα, αλλά σε σχέση με το πόσο, έχει, πόσο έχουν υποθεί για αυτό το ψήφισμα, ε, Τελικά οι πόροι που διατίθενται για την ειρήνη και την ασφάλεια, μόλι 2% αυτών των πόρων έχουν να κάνουν με το να προχωρήσει το ζήτημα αυτό. Λιγότερο από 2%. Λοιπόν, τελικά αυτέ οι ειρηνευτικέ διαδικασίες ε, ε, το αποτυπώνουν αυτό. Εδώ βλέπετε μία μελέτη που είναι ίσως ε, και η πιο πλήρης όπου βλέπουμε το ρόλο των γυναικών στις ε, μεγάλες ερνευτικές διαδικασίες εδώ και 20 χρόνια περίπου και βλέπετε εδώ είναι αρκετά ζωφερή η εικόνα, λιγότερο από 2% των επικεφαλής διαμεσολαβητών, 4% όλων όσων ε, έχουν υπογράψει τις συμφωνίες και μόλις και λιγότερο από 10% όσων συμμετέχουν γενικότερα στα τραπέζι διαπραγματεύσεων που συζητούν δηλαδή ε, για τα ζητήματα αυτά. λιγότερα από 10%. Οπότε, όπως βλέπετε, είμαστε αρκετά μακριά από τους ε, στόχους που είχαμε θέσει. Πώς το βλέπουμε τώρα εμείς, ε, με βάση την πραγματικότητα επιτόπου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το θετικό είναι ότι αυτό το πλαίσιο έχει θέσει το ζήτημα επιτάπητος. Ε, στο παρελθόν κανείς δεν ρωτούσε πού είναι οι γυναίκες στην ελληνική διαδικασία. Είναι και αυτό ένα σημείο αφετηρίας. Είναι μια αρχή ε, να γνωρίζουμε τουλάχιστον την απουσία του. Όμω, ό,τι αφορά το ποιο συμμετέχει στι διαπραγματεύσει αυτέ, ε, ποιε είναι οι επίσημε διαδικασίε, εκεί βλέπουμε ότι είναι πολύ λίγε οι γυναίκε. Το έδειξαν οι τα προηγούμενα στατιστικά. Το βλέπουμε στην ειρηνική διαδικασία στην Ιεμένη, στη Συρία. Δεν υπάρχουν πολλέ γυναίκε εκεί. Όμω, πρέπει να πω ότι όταν, όταν μιλάμε για ειρηνευτικέ διαδικασίε σε άλλα επίπεδα, όχι στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο απαραίτητα, αλλά σε τοπικό επίπεδο, ε, δημιουργία, οικοδόμηση εμπιστοσύνη, εκεί οι γυναίκε παίζουν ένα πολύ πιο σημαντικό ρόλο. Στην Ουκρανία ε, μπορούμε να μιλήσουμε και για ε, μια πιο θηλυκή κοινωνία των πολιτών. Βεβαίω είναι ζητήματα που θεωρούνται λιγότερο σημαντικά από πολιτική πλευρά, ε, δεν πρέπει να χαθούν όμως και αυτές οι ευκαιρίες. Γιατί λοιπόν συμβαίνει αυτό, ποια είναι τα εμπόδια. Ενώ υποτίθεται ότι όλοι δεσμευόμαστε προς μια κατεύθυνση, τα στατιστικά μας λένε τα αποτελέσματα είναι τα αντίθετα. Μπορούμε να αναφερθούμε εδώ σε μια σειρά από λόγους. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια γενικότερη πρόκληση ό,τι αφορά τη διαμεσολάβηση και το διάλογο. Ε, είναι πολύ λιγότερο το πεδίο ε, στην διαμεσολάβηση αυτή, πολύ μικρότερο ε, για τη διαμεσολάβηση γενικότερα και για την κοινωνία των πολιτών και αυτό ε, παρεμποδίζει και τη συμμετοχή των γυναικών. Το CMI πέρσι οργάνωσε μια σειρά από συναντήσεις με ακαδημαϊκούς, με ανθρώπου που έχουν συμμετάσχει στι διαπραγματεύσει ή που έχουν παίξει ρόλο του μεσολαβητή και προσπάθησε να εντοπίσει πού βρίσκεται το πρόβλημα. Και έφτασε στο συμπέρασμα ότι είναι θέμα ε, πραγματικά αντίληψη. Ε, υπάρχουν κάποια εμπόδια δηλαδή στο μυαλό μα. Είναι κάποιοι μύθοι οι οποίοι εξακολουθούν ε, να επιβάλλονται ε, σε ό,τι αφορά τα, τη μεσολαβηση Κάποιοι μιλάνε για ζητήματα που αφορούν γυναίκες, ζητήματα γυναικεία. Τι θα πει αυτό. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την ειρήνη και την ασφάλεια που δεν αφορούν τις γυναίκες. Επίσης, ε, ε, ουσιαστικά αρχίζουμε να εξετάζουμε το θέμα της, του διαλόγου ε, όταν ξεκινούν διαπραγματεύσει, χωρίς να, να το εξετάσουμε όταν θεσπίζεται η ατζέντα. Βεβαίω υπάρχουν πλέον σύμβουλοι για ζητήματα φύλου, αλλά αυτοί βρίσκονται ε, στην αρχή Επίσης, ε, συνήθως οι γυναίκες παρουσιάζονται ως φωνές και όχι ως πραγματικοί πολιτικοί παράγοντες. Δηλαδή απλά ακούμε την άποψή τους, χωρίς όμως ε, αυτές οι απόψεις να είναι δεσμευτικές για την ε, ειρηνευτική διαδικασία. Δηλαδή δίνει μια εντύπωση ότι η δημοσιολάβηση αφορά κάποιους ε, άντρες που καπνίζουν, πίνουν ουίσκι και συζητούν και καταφέρνουν να βρουν μια λύση. Υπάρχει και ένας μύθος ότι ζητούνται περισσότερα απολυτικά στοιχεία για την συνεισφορά των γυναικών. Έχουν γίνει μελέτες γι' αυτό που αποδεικνύουν ότι υπάρχει ένας σχετισμός, αλλά θεωρούμε ότι το, λάθος, το, το ερώτημα από την αρχή είναι λάθος. Γιατί να ρωτήσει κανείς, να ζητήσει κανείς στοιχεία, γιατί το ζητάμε αυτό για τους άντρες. Οι πρώτε προσπάθειε για τη συμμετοχή των γυναικών λοιπόν έχουν έρθει πολύ αργά, είναι ad hoc και είναι απομονωμένε από την υπόλοιπη ειρηνευτική διαδικασία. Τι μπορεί να γίνει γι' αυτό, πολύ σύντομα. Υπάρχουν και εργασίε αυτή τη Επιτροπή. Ε, μακροπρόθεσμη επένδυση. Δεν περιμένουμε δηλαδή, να ξεκινήσει μια σύραξη ή μια ειρηνευτική διαδικασία. Προσπαθούμε ήδη να επενδύσουμε σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό επίπεδο, έτσι ώστε οι γυναίκε να έχουν μεγαλύτερη ε, δύναμη ε, από την αρχή. Τώρα υπάρχουν τέσσερις πτυχές ε, για το τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει τα λόγια μας να τα συνοδεύουμε με συγκεκριμένους πόρους. Αυτό το 2% είναι πραγματικά ατιμωτικό, πρέπει η Ευρώπη να το αλλάξει αυτό, να δώσει το καλό παράδειγμα. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε ε, τοπικούς τρόπους ε, ε, ενίσχυση των γυναικών σε αυτές τις διαδικασίες. Συχνά προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιε διεθνείς συνταγέ, οι οποίες όμως δεν ταιριάζουν πάντα σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει να ακούσουμε τους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς, να δούμε ποιε είναι οι πραγματικές ανάγκες τους. Τρίτον, πρέπει ε, να, να συνδυαστεί με τη διαμεσολάβηση η ατζέντα των Ηνωμένων Αθνών. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να οδηγήσει μια συνέργεια. Και τέλος, συχνά ακούω από τι γυναίκε ε, στι χώρε σύραξη ότι ζητούν πρόσβαση. Το πρώτο που ζητούν είναι πρόσβαση και το μόνο. Ε, όταν έχουν πρόσβαση μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν. Μπορούν να ανοίξουν κάποιες πόρτες, μπορούν να κάνουν να ακουστούν κάποιες φωνές ε, σε αυτή την πολιτική συζήτηση. Αυτά είχα να πω εγώ εισαγωγικά. Αναμένω τη συζήτηση. Σας ε, ευχαριστούμε πολύ. Ε, κυρία Ποτάνεν, πριν δώσω το λόγο στην κυρία Μαγκαγιώνα, θα ήθελα να καλωσορίσω μια ομάδα ε, που έχει, επισκεπτών που έχει φέρει η κυρία Νόιχελ από το SPD. Η κυρία Μαγκαγιόν λοιπόν έχει το λόγο, είναι ερευνήτρια ε, της ε, Διεθνούς ε, Ομοσπονδίας για την Ειρήνη και την Ελευθερία. Θα μιλήσω στα Ισπανικά για την ημιτρική μου γλώσσα. Λοιπόν, αποδέχτηκα την πρόσκληση γιατί ήθελα να αναφερθώ εδώ μπροστά σας ε, σε δύο θέματα, δύο περιπτώσεις στην Κολομβία και τη Δυτική Σαχάρα για θέματα τα οποία είναι θέματα που σχετίζονται με, με αυτά που σας απασχολούν. Πρόκειται για δύο φορά πολύ σημαντικά, ε, στα οποία συμμετέχουν οι γυναίκες σε ειρηνευτικές διαδικασίες ε, και είναι σημαντικό να μην τις αφήσουμε μόνες, να τις υποστηρίξουμε. Όπως ε, είπε προηγουμένως ε, και η ομιλήτρια που μίλησε πριν από μένα, είναι σαφές πλέον μέσω και πολλών τεκμηριωμένων ε, μελετών ότι οι γυναίκες όταν συμμετέχουν σε ειρηνευτικές διαδικασίες ε, έχουν πολύ θετικό αντίκτυπο και μάλιστα ε, αυτό έχει αποδειχθεί και μέσα από διαφορετικά μοντέλα συμμετοχής. Δηλαδή μπορεί κανείς με διάφορους τρόπους να συμμετάσχει σε αυτήν την διαδικασία και να έχει καλά αποτελέσματα όχι μόνο σε ποσοτικό αλλά και σε ποιοτικό επίπεδο. Ε, και ο αντίκτυπος των ε, γυναικών ε, στην επίτευξη της ειρήνης. Σχετικά με αυτό αναφερόμαστε στην διάρκεια της ειρήνης ε, και ε, αναφέρεται ότι μια συμφωνία ε, μπορεί κατά 35% περισσότερο να διαρκέσει εάν έχουν συμμετάσχει γυναίκες σε αυτήν την διαδικασία. Και όταν η Αλεξάνδρα Μπουκέτε αναφέρεται στην πολιτική των γυναικών, απαντά η πολιτική των γυναικών είναι η πολιτική, δηλαδή το, το σύνολο. Και δεν θα μπούμε σε μια γωνίτσα της πολιτικής, το ίδιο, ε, στο ίδιο ε, ε, καταλήγει η μελέτη αυτή όσον αφορά τα επιτεύγματα των γυναικών όταν συμμετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, πολλές μελέτες όπου οι διαδικασίες ειρήνευσης ξεπερνούν κατά πολύ την απλή κατάπαυση του πυρός ε, και μπορούν να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της κοινωνίας μετά από το τέλος ε, της ε, σύραξης. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ συγκεκριμένα στην περίπτωση της Κολομβίας. Γνωρίζετε ότι η ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία ήταν μία από τις μακρότερες που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Να σας πω ότι το 2008 ε, η εθνική ομάδα συμφιλίωσης με προσκάλεσε και ήμουν ε, σε μια στρογγυλή τράπεζα ε, με 11 άνδρες. Είχαμε μονάχα μία εκπρόσωπο εκτός από μένα που με είχε καλέσει η Ισπανική Πρεσβεία για να μιλήσω για το θέμα αυτό. Είχαμε και μία γυναίκα εκπρόσωπο των θυμάτων. Από αυτή τη στιγμή μέχρι την επίτευξη των συμφωνιών, οι διαδικασίες που ακολούθησαν οι γυναίκες στην ε, ε, Κολομβία ήταν πραγματικά υποδειγματικές κατάφεραν να προωθήσουν και να ε, τις ε, συμφωνίες τους, τις ιδέες τους, να τις υποστηρίξουν ε, η διεθνής κοινότητα και άλλοι, ε, να δημιουργήσουν ε, διάφορες οργανώσεις όπως ας πούμε η, Οδός της Ειρήνης των Γυναικών της Κολομβίας κλπ. Και κατάφεραν λοιπόν να διεκδικήσουν την συμμετοχή τους στις ειρηνευτικές διαδικασίες μέσα από μια υποεπιτροπή ε, ισότητας των φύλων και κατάφεραν με τον τρόπο αυτό ε, να δώσουν μια πιο ε, συγκεκριμένη συμβολή στις ειρηνευτικές διαδικασίες. Πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλέ οι γυναικείες οργανώσεις οι οποίες εργάστηκαν προς την κατεύθυνση αυτή και επίσης ε, οι γυναίκες των Ηνωμένων Εθνών ε, και λοιπά ε, συνέβαλαν στην διαδικασία. Επίσης, οι γυναίκες κατάφεραν να συγκαλέσουν δύο διασκέψεις κορυφής ε, οι οποίες ε, δεν προχώρησαν μόναχα σε συμφωνίες αλλά ε, έδωσαν και μία έντονη παρουσία των γυναικών σε αυτές τις εθνικές διασκέψεις κορυφής ακριβώς οι γυναίκες έδωσαν το στίγμα τους πριν από αυτό. Υπήρχαν μελέτες όπως ας πούμε η αλήθεια των γυναικών που οδήγησε και στην δημιουργία της λεγόμενης Ρούτα Παθήφικα Μουχέρες», την ε, ειρηνευτική οδό των ε, γυναικών ε, και επίσης την συμμετοχή των γυναικών θυμάτων. Πραγματικά ήταν μια υποδειγματική μελέτη η οποία ελήφθη υπόψη από την Επιτροπή για την Αλήθεια στην Κολομβία. και ε, η Άγχελα ε, Σαλαφάρ ε, ήταν η οποία ήταν η εκπρόσωπος των γυναικών στην Επιτροπή αυτή. Τώρα, γιατί θέλω εδώ να αναφέρω αυτήν την περίπτωση. Το κάνω γιατί οι συμφωνίες ε, ε, που επετεύχθησαν ε, για την ειρήνη αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κίνδυνο. Η παρούσα κυβέρνηση αντιτίθεται σε αυτές τις ειρηνευτικές διαδικασίες και να σας πω ότι πριν από ένα μήνα ο πρόεδρος της Κολομβίας ε, ανακοίνωσε ότι αντιτίθεται σε έξι άρθρα ε, της ειδική Επιτροπής ε, για την Αλήθεια και η Πατρίθια Λινάρες είπε ότι οπωσδήποτε θα αντιταχθούμε σε αυτό. Είναι σημαντικό γιατί εδώ έχουμε νομολογία που αφορά την ειρήνη και επομένως οτιδήποτε θέτει σε κίνδυνο την νομολογία αυτή θέτει σε κίνδυνο την ε, ειρηνευτική διαδικασία ε, και η διεθνής κοινότητα ε, πήρε μέρος σε αυτές τις διαδικασίες ειρήνευσης και επομένως αυτήν την συμφωνία. Άρα εδώ τίθεται ένα αμφιβόλο η ίδια η αξιοπιστία της διεθνούς κοινότητας. Δεν πρέπει να αφήσουμε μόνη της την χώρα. Εδώ βλέπετε μία εικόνα από απομακρυσμένη περιοχή ε, όταν μιλάμε για τέτοιες περιοχές στην Κολομβία είναι πραγματικά απομακρυσμένες. Πρέπει κανείς να διασχίσει ε, βουνά, χυμάρους, ποτάμια κλπ. για να φτάσει σε αυτά τα απομακρυσμένα μέρη. Ε, και εδώ οι άνθρωποι που βλέπετε μας ζήτησαν να μην τους αφήσουμε μόνους τους. Επομένως, εγώ έρχομαι εδώ για να μιλήσω εξ ονόματός τους. Είμαι η φωνή τους αυτή τη στιγμή έτσι ώστε να συνεχίσει η διεθνής ε, κοινότητα να εργάζεται ε, ε, έτσι ώστε η Κολοβιανή κυβέρνηση να μην αναθεωρήσει αυτές τις συμφωνίες. Εμείς επισκεφθήκαμε και κάποια μέρη στα οποία ζουν οι παλιοί αντάρτες των ΦΑΡΚ και πραγματικά αυτή, αυτή τη στιγμή ε, διανύουν περίοδο μεγάλης νομικής ε, ανασφάλειας. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Πιστεύω ότι θα πρέπει ε, Ε, είχαμε, ήρθαμε σε επαφή και με τους LLN ε, και ε, βλέπουμε ότι έχουν μεγάλο προβληματισμό σε σχέση με τα όσα αρχίζει η κυβέρνηση να κάνει σε σχέση με τους φάρκα. Εμείς ε, ως Ευρωπαϊκό Τμήμα της Will Europa ε, κάνουμε αυτήν την ε, προσπάθεια, αλλά θέλω να προχωρήσω με ταχύτητα και να περάσω στο επόμενο παραδειγμά μου που είναι αυτό της Δυτικής Σαχάρας. Πρόκειται για εδάφη τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία από απικιοποίησης. Οι άνθρωποι αυτοί, οι πολίτες της Σαχάρας ζουν στρατόπεδα προσφύγων από το 1975 και από όταν έπεσε η δικτατορία στην ε, ε, Ισπανία και υπάρχει, υπάρχουν βέβαια και τα κατεχόμενα από το Μαρόκο εδάφη. Εμείς ε, ήρθαμε σε επαφή και συμμετείχαμε στις διαδικασίες των συζητήσεων που ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 2018. Οι γυναίκες έχουν έχουν ε, προχωρήσει στην αποστολή μιας επιστολής την οποία προσυπογράφουν 50 ανεξάρτητες ε, γυναίκες ε, Σαχαράουι και που αναφέρουν ακριβώς τα προβλήματα και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να προωθηθεί η ειρηνευτική διαδικασία. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτές τις γυναίκες που οικοδομούν την ειρήνη εάν διευρύνουμε τη φωνή τους, εάν μπορέσουμε να κάνουμε πιο ορατή την γενεολογία ε, ε, που έχουν ε, οι γυναίκες στην ιστορία των ειρηνευτικών διαδικασιών. Κοιτάξτε, εμείς μιλάμε για την βία κατά των γυναικών, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για τις γυναίκες ενάντια στη βία. Ο Νιούτον είπε, ο φυσικός είπε ότι έχουμε την δυνατότητα να φτάσουμε πάρα πολύ μακριά στην ε, επιστήμη γιατί βασιζόμαστε σε πλάτες ε, γιγάντων. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε και εμείς γιατί οι γίγαντές μας είναι αυτές οι γυναίκες οι οποίες σε βάθος χρόνου ε, έχουν οικοδομήσει την ειρήνη. Αυτό είναι ένα μεγάλο κληροδότημα, είναι ένα κληροδότημα γυναικών, φιλοσόφων, δημιουργών, ε, ε, γυναικών που ε, κάνουν την καινοτομία. Οι ειρηνευτικές, οι, οι για την ειρήνη δημιουργήθηκαν σαν κίνημα στη Χάγη το, το 1915. Ε, και πραγματικά ξεκίνησε ήδη μια μεγάλη διαδικασία η οποία καταλήγει πάντα στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να υπάρχει μέλλον εάν δεν υπάρχει ειρήνη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μαγκαγιόν. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Λάουρα Ντάβις. η οποία προέρχεται από το European Peace Building Liaison Office. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, και μέλη της Επιτροπής. Μιλάει εκ του Γραφείου για την ειρήνευση, μια υπηρεσία που έχει παγκόσμια δράση εδώ και πολλά χρόνια για την οικοδόμηση της ειρήνης και την αποτροπή συγκρούσεων. Την προηγούμενη Παρασκευή οργανώσαμε έναν συνεδρίαση από με την ΕΠΛΟ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία συναντήθηκαν 15 μεσολαβήτριες γυναίκες από τη Βόρεια Αφρική, το τη Αφρική, την Ιεμένη, την Ουκρανία και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και δικά μας μέλη για την διχείριση κρίσεων, για να ξεπεράσουμε τα στερεότυπα και να δούμε πώ μπορούν, πώς μπορεί η να υποστηρίξει τι γυναίκε διαμεσολαβητρίε, Θέλω να πω ότι οι γυναίκε οι οποίες εμπλέκονται στην διαμεσολάβηση και όχι στο ευρύτερο πλαίσιο της ειρήνευσης. Ε, και για να το αυτό υπάρχουν δύο παρεμβάσεις ε, που γίνανε και από την Κάρμεν και από την Ιωάννα πριν από μένα. Μια μεγάλη σημαντική μαρτυρία από μια από αυτές τις γυναίκες που ε, πλάκησε θέματα τέτοια στη βάση είναι το πώς γίνεται η διαμεσολάβηση από τις γυναίκες, πώς ε, δεν αναγνωρίζεται δημόσια. Άρα θα πρέπει το Κοινοβούλιο να αναγνωρίσει την προσπάθεια των γυναικών να τις φέρει στην δημοσιότητα. Μία από αυτές οι οποίες σχολείς είπε ότι απλά βγήκαμε έξω και κάναμε ό,τι χρειάστηκε να κάνουμε. Και μετά καταλαβαίνω ότι αυτό που κάναμε ήταν η διαμεσολάβηση. Και αυτό μας φαίνεται ένα δεύτερο σημείο που πολύ συχνά έχουμε πολύ ξεπερασμένε απόψει για το τι είναι η διαμεσολάβηση. Και αυτοί οι ορισμοί πολύ συχνά παραβλέπουν το έργο που κάνουν οι γυναίκε στι κοινότητε για την ειρήνευση και για την διάσωση ζωών. Κάποιες άλλες μαρτυρίες από τις συμμετέχουσες έκαναν λόγο για την σημασία του ρόλου των φίλων στην κοινωνία. Η Ιωάννα μίλησε για τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και να επανέλθω σε σχόλια που έκαναν, τα οποία παρουσιάσαμε στην είπατε εκπρόσωπο χθε. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι πώς οι γυναίκες δημοσιογραφητρίες περιγράφουν τον εαυτό τους ως δυνατές μέσα στην αδυναμία τους. Σε καταστάσεις σύγκρουσης όπου οι άντρες έχουν δυσκολία να βρουν σημεία για να παρέχουν μαρτυρίες και πολλές φορές οι γυναίκες είναι αυτές που θα πάνε σε αυτά τα σημεία για να μιλήσουν Οι συγκρούσει είναι θέμα των αντρών. Οι γυναίκε αποκλείονται από αυτό. Δεν θεωρούνται σημαντικέ σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή, αυτός ο αποκλεισμός είναι πιο ισχυρός ε, στις ε, συμφωνίες. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουν κατά νου οι παρατηρητέ σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα βλέπουμε ότι εκεί που εμπλέκονται σε διαδικασίες γυναίκες διαμεσολαβητρίες μπορούν να επιφέρουν με διαφορετική διάσταση για τις ανάγκες της κοινωνίας και για αυτό που συμβαίνει στη βάση. Και αυτό ε, σημαίνει ότι υπάρχει μία έννοια ασφάλειας και διαφέρουν ε, οι διαδικασίες γενικότερα όταν σε αυτές, ε, από, από, όταν σε αυτές συμμετέχουν μονάχα τύπους που συμμετέχουν και εμπλέκονται στην σύραξη. Οι γυναίκες που εργάζονται στην Ιεμένη κάνουν λόγο για περιοχές ε, όπου έχουν πιο πολλή εξουσία. Αυτό πολλές φορές το παραβλέπουν οι ξένοι παρατηρητές και ήδη γίνεται διαμεσολάβηση σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου όπου οι γυναίκες έχουν ηγετικό ρόλο. Από την άλλη πλευρά η Ιωάννα έκανε αναφορά σε αυτό ότι σε χώρες όπως την Ουκρανία η διαμεσολάβηση είναι αποκλειστικά έργο των γυναικών επειδή είναι μια εργασία πολύ χαμηλά αμοιβόμενη. Και πολλές φορές θεωρείται ότι είναι χόμπι και όχι πραγματικό έργο ε, που προσφέρει και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης ένα από τα πράγματα που ισχύουν σε πολλά μέρη είναι η απειλή και ο εκφοβισμός που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διαμεσολαβήτριες. Επιπρόσθετα έχουν και απειλές σε σχέση με την ασφάλειά τους, αλλά αποτελούν και στόχο για άλλες, ε, ε άλλου εκφοβισμού φόβο ότι θα τις δυσφημίσουν στην κοινότητά τους και στις οικογένειές τους για το έργο που προσφέρουν. Και μία από, την, μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πώς αυτές οι γυναίκες και πώς η εικόνα των γυναικών διαμεσολαβητών διαστρεβλώνεται και δημιουργεί κινδύνους και για τις γυναίκες και για τις ε, οικογένειές τους και πλέον για τις κοινότητές τους είναι μια άλλη μορφή επιτυχημένη οικοδόμησης ειρήνη. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται οικοδόμηση εμπιστοσύνη σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Και αυτό είναι πιο πιθανό να συμβεί με τη συμμετοχή γυναικών περισσότερο παρά Είχε ένα πολύ ωραίο κόμικ η Ιωάννα Και αυτό που πρέπει να αναγνωρίσουμε, ότι ανεξάρτητα με την προέλευση των ε, γυναικών διαμεσολαβητών, έχουν πάρα πολλές ε, ευθύνες και πρέπει να είναι διαθέσιμες ανα πάσα στιγμή για να μπορούν να προσφέρουν ε, το έργο τους. Παράλληλα έχουν και την ευθύνη απέναντι στην οικογένειά τους και στους εργοδότες τους. Άρα, ο χρόνος των συνεδριάσεων, των συζητήσεων, γίνονται πολύ συχνά το βράδυ, αργά, που είναι πολύ δύσκολο για τις γυναίκες ε, να παρακολουθήσουν και να παρευρεθούν. Θα ήθελα λοιπόν να ολοκληρώσω με κάποιες συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα πιο ευρέως, να σχολιάσω αρχικά τη στρατηγική ε, προσέγγιση της Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συμπέρασματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, στα οποία ε, συμμετείχαμε γιατί, και χαιρόμαστε γιατί ενισχύουμε τη συμμετοχή ε, των γυναικών στις δικασίες αυτές. Όσον αφορά τις πολιτικές που συνδέονται με το 1325 Αν υπομονούμε να δούμε την ε, εφαρμογή αυτού του σχέδιου δράσης από όλα τα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην εξωτερική και στην εσωτερική δάση και ελπίζουμε ότι αυτή η Επιτροπή θα διδραματίσει σημαντικό ρόλο για να διασφαλίσει ότι θα εφαρμοστεί όντως αυτό το σχέδιο δράσης. Κάποιες από αυτές τις στοιχείες εμφανίζονται και στο σχέδιο του προγράμματος δράσης και στη στρατηγική προσέγγιση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, αποτρέψει τους αποκλεισμούς και σε όλα τα παιδά και στην διπλωματία θα πρέπει η συμπερίληψη γυναικών να αυξηθεί γιατί δεν είναι απαρκή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δημιουργήσει ε, ομάδες που θα συμπεριλαμβάνουν και γυναίκες για δύο λόγους. Πρώτον, είναι πολύ πιθανό να βελτιωθεί η ποιότητα της ομάδας, αλλά επίσης, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκτήσει μεγαλύτερη αξιοπιστία Και το δεύτερο σημείο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πάρα πολλέ ε, επιτροπέ και διαλόγου και διαδικασίε σε παγκόσμιο επίπεδο και σε διπλωματικό επίπεδο, ακόμα και σε επίπεδο ε, εντό των κοινοτήτων και γι' αυτό θα πρέπει να απαιτήσει για τη συμμετοχή κατά 30% των γυναικών να τηρηθεί από όλα από όλου του συμμετέχοντες. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει τη δικτύωση και την κατάρτιση διαμεσολαβητών και γυναικών και αντρών και να συνδέσει τι γυναίκες με διάφορες ευκαιρίε. γιατί οι γυναίκες δεν ναι, μπορεί να είναι αρκετά καταρτισμένες αλλά να μην έχουν τις σωστέ διασυνδέσει ε, για να εργαστούν στη διαμεσολάβηση ως κοινωνία πολιτών και σε όλες τις μορφές διαδικασιών ειρήνευσης είναι πολύ βασικό να υπάρχει μια ανάλυση για τα φύλλα. Γιατί όταν κάνουμε λόγο για ανθρώπους, κάνουμε λόγο για το φύλλο τους. Και δεν υπάρχουν ειρηνευτικές διαδικασίες που θα είναι αποτελεσματικές αν αποκλείουν από την διαδικασία κάποιες πολύ σημαντικέ στοιχείες τη κοινωνία. Όλα αυτά θα πρέπει να τηρηθούν και στο σχέδιο δράσης και να εφαρμοστούν. Και τέλος, κάποιες ακόμα σκέψεις, η διαμεσολάβηση είναι πολύ επιβαρυντική και για την ε, φυσική, σωματική υγεία και για την πνευματική υγεία των γυναικών θα πρέπει να παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αποκατάσταση για τις γυναίκες που συμμετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες. Είναι μια πρακτική η οποία έχει πολύ σκληρές επιπτώσεις σε αυτούς που συμμετέχουν. Ο ρόλος των γυναικών και των αντρών σε περιοχές συγκρούσεων, σειράξεων και η παρουσίασή τους στα μέσα μας και στην ενημέρωση μπορεί να αλλάξει τα προτεραιότητα, άρα θα πρέπει να στηρίξουμε project στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να δείξουμε πώς έχει κατάσταση. Επίσης, η συμπερίληψη γυναικών ε, σε ομάδες υψηλού επίπεδου είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι επίσης κάτι που θα πρέπει να στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, να αναφερθώ σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι θα πρέπει να υπάρξει δημόσια αναγνώριση των γυναικών διαμεσολαβητριών. Είναι πολύ τιμή η δουλειά τους, αλλά η δουλειά τους αυτή παραβλέπεται. Γι' αυτό θα ήθελα να παροτρύνω την Επιτροπή αυτή να αναγνωρίσει το έργο των γυναικών αυτών και να ρίξει το φως πάνω στο έργο τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα η Κατρίνα Κρουχόβνα του, Κέντρου Ειρήνης Κατά Καταπολέμησης της Βίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να μιλήσω μαζί σας και να ανταλλάξω ε, απόψεις ε, για την ε, οικοδόμηση μιας κουλτούρας ειρήνης και το ρόλο των γυναικών σε αυτήν την οικοδόμηση. Είμαστε κάπου μεταξύ απελπισίας και ελπίδας. Εγώ προέρχομαι από την Κροατία και θα σας μιλήσω κυρίως ε, για τη δική μου εμπειρία. Στη συμμετοχή μου στην εμπόλεμη κατάσταση στην Κροατία και βεβαίως στην οικοδόμηση της ειρήνης στη συνέχεια. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Κροατία Έτσι και τώρα ζούμε σε βία εποχή. Και αναρωτιέμαι, όπως αναρωτιόμουν πριν από 20-25 χρόνια, μπορεί η μη βία να υπερνικήσει τη βία. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αναρωτηθούμε. Ε, να ρωτήσουμε τον εαυτό μας ως πολίτες, Το λέω και ω πολίτη βεβαίω μια χώρα των Δυτικών Βαλκανίων, τη Κροατία, που έζησε, ζήσαμε στη δική μας εποχή τον πόλεμο και τη βία που φέρνει. Δεν είναι ένα καινούριο ζήτημα όμως. Είναι μία αρχή πάνω στην οποία βάσισαν την ε, δεσμευσή τους οι πολλές γυναίκες που έδωσαν αυτή τη μάχη. Από την δεκαετία του 1990 προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για την δημιουργία ειρηνικών σχέσεων και μέσα στον πόλεμο. Τώρα, 20 χρόνια αργότερα, εξακολουθούμε να σκεφτόμαστε στην περιοχή μας, στην Κροατία και στην Ευρώπη πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε αυτές τις ειρηνικές σχέσεις. Η ιστορία της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μας είναι πηγή έμπνευση. Είναι η ελπίδα ε, μιας ειρηνευτικής, ε, μιας ειρηνικής μάλλον ε, ένωσης. Στη δική μου διαδρομή έχω την τιμή να συνεργάζομαι με πολλές και διαφορετικές γυναίκες αυτές που δραστηριοποιούνται σε ειρηνικά κινήματα, φεμινιστικά, οικολογικά. Ε, σε αυτές που προσπαθούν να προωθήσουν το διάλογο μεταξύ των θρησκειών ε, για να προωθήσουν έτσι τη δικαιοσύνη και την ειρήνη. Οι ακτιβισμοί αυτοί διαφέρουν γίνεται, υπάρχουν πολύ ισχυρά αντιπολεμικά ε, κινήματα όπως οι γυναίκες με τα μαύρα στη Σερβία ε, αλλά υπάρχουν και πιο αόρατα ε, αυθόρμητα κινήματα σε τοπικές κοινωνίες για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης. Έμαθα πολύ επίσης για το ρόλο των καθηγητών, των δασκάλων στα σχολεία, στις ε, τοπικές κοινωνίες. Οι γυναίκες οι ακτιβιστές ειρηνιστές εξετάζουν ακόμα και σήμερα πώς να αντιμετωπίσουν τα αισθήματα του παρελθόντος, τι γίνεται με τα δικαιώματα των θυμάτων ε, ή των επιζώντων που έχουν επιστεί βιασμούς ενδεχομένως, τι συμβαίνει με τους αγνοούμενους. Υπάρχει μια νέα γενιά γυναικών σήμερα που συμμετέχει σε αυτούς τους πολιτικούς αγώνες κατά των πολλαπλών μορφών βίας και στην περιοχή μας αυτό είναι πιο έντονο λόγω του πολέμου, λόγω της μεταπολεμικής αυτής κατάστασης. Κατά τη διάρκεια του πολέμου και τα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο, στην περιοχή από όπου προέρχομαι, ο πόλεμος ε, ε, δίχασε την κοινωνία μας τόσο γρήγορα που δεν μπορέσαμε καν να δημιουργήσουμε μια κοινή πλατφόρμα, κάποιο ειρηνευτικό κίνημα. Έτσι λοιπόν τα όποια κινήματα κινήθηκαν παράλληλα και ξεχωριστά. Όμως η συνεισφορά μας στην οικοδόμηση της ειρήνης ε, ήταν ότι βρήκαμε, βρήκαμε έναν τρόπο παρόλα αυτά να ανοίξουμε ένα διάβλο επικοινωνίας, να την ενισχύσουμε ε, να συνεργαστούμε μέσω δικτύωσης στην περιοχή και είχαμε και ακόμα έχουμε περιφερειακές δραστηριότητες όπως η πρωτοβουλία της Περιφερειακής Επιτροπής για την ε, αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τα θύματα του πολέμου. Βεβαίως, παρόλα αυτά, τον πόλεμο δεν το σταματήσαμε. Ούτε επηρεάσαμε την έκβασή του. Όμως, η συνεισφορά μας στην ειρήνη Ξέρετε, η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ακτιβιστών είναι γυναίκες ήταν η δημιουργία κάποιων αξιών βάσει των οποίων μια δημοκρατική κοινωνία μπορεί να αναπτυχθεί. Και οι προσπάθειες οικοδόμησης της ειρήνης στην περιοχή έχουν παίξει αυτό το ρόλο. Διότι είναι απαραίτητο σήμερα. Υπάρχει ανάγκη να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να σώσουμε και να προωθήσουμε και το ευρωπαϊκό ε, ειρηνικό όραμα αλλά και να προλάβουμε ε, ενδεχόμενες σειράξεις σε περιοχές ε, όπου ελοχεύουν κίνδυνοι στο Κοσφοπέδιο, στη Βοσνία, στη Μακεδονία Όμως δεν το σκέφτομαι σήμερα. Βλέπω ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες με αυτό που γινόταν κατά τη του πολέμου, αλλά και με τα πολεμικά. Και ψάχνω απελπισμένα ξανά την ελπίδα. Νομίζω ότι και στην Ευρώπη τα ίδια ζητήματα τίθενται. Τα ίδια πράγματα έχουμε να σκεφτούμε. και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία που μου δίνουν ελπίδα. Θα σας πω ποιοι είναι οι δύο πυλώνες αυτής της ελπίδας για μένα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει παγκόσμια κατάσταση. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι υπάρχει μια κοινή παγκόσμια αναγνώριση της ανάγκης ειρηνικών κοινωνιών. Είναι ένας ε, ένα, ένα στόχος ε, της βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς ειρήνη, ε, λέει η σχετική διακήρυξη. Και δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς βιώσιμη ανάπτυξη. Στο άρθρο 4, 7, γίνεται λόγος ε, για την εκπαίδευση σε ό,τι αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη, την ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των δύο φύλων, την προώθηση μιας κουλτούρας ε, ειρήνης, μη βίας και πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας ε, επιβεβαιώνει ότι η πρόληψη λειτουργεί, πιάνει τόπο. Δηλαδή αυτά που γίνονται μέσω οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, μέσω της εκπαίδευσης, μέσω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δύο φύλων, τη δημοκρατική συμμετοχή, την αλληλοκατανόηση, την ανοχή, την ελεύθερη ροή πληροφοριών. Όλα αυτά δημιουργούν μια κουλτούρα ειρήνης. Και βεβαίως ας επανέλθουμε τώρα στο κοινωνικό επίπεδο. Πρέπει να συναντήσουμε τις γυναίκες εκεί που βρίσκονται Το άλλος πυλώνας λοιπόν για μένα, για την ελπίδα μου, είναι η εμπειρία που έχω μέσα μου και που έχω αποκομίσει από τον πόλεμο. Ήμουν από τους ιδρυτές ε, του κέντρου ειρήνης μη βίας ε, στην Κροατία, ε, μέσω πολέμου και η εμπειρία μου λέει ότι μπορεί κανείς να οικοδομήσει την ειρήνη, να την προετοιμάσει, ενώ, ενώ λαμβάνει χώρα πόλεμος. Και λέω ότι αυτό πρέπει να το έχουμε κατά και εμείς στην Ευρώπη σήμερα. Πώς συνέβη αυτό. Μια μικρή ομάδα ανθρώπων, πλειοψηφία εκ των οποίων ήταν γυναίκες, άρχισαν να σκέφτονται πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο. Πρέπει να τον προλάβουμε και πολύ γρήγορα διαπιστώσαμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε. <coughs> Δεν εξαρτάται από εμά. Όμω αξίζει να σκεφτόμαστε τότε κάτι άλλο. Τι είδου κοινωνία θέλουμε να έχουμε μετά τον πόλεμο, στο μέλλον. Και μιλούσαμε γι' αυτό δύο μήνες και φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι θέλουμε μια κοινωνία που να είναι πιο ανθεκτική στη βία που να έχει μεγαλύτερες δυνατότητες μη βίας ε, και μη βίαιης επίλυσης των διαφορών και των αδικιών. Ορίσαμε λοιπόν τη βιώσιμη ειρήνη ως ένα, μια δυναμική κατάσταση διαρκούς ανοικοδόμησης, βελτίωσης των σχέσεων για μεγαλύτερη δικαιοσύνη, μεγαλύτερη συμπερίληψη, συνεργασία και αλληλεγγύη στο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο. Ήταν λοιπόν αυτό ένα όραμα μιας κουλτούρας ειρήνης. Ανάπτυξης μιας κουλτούρας ειρήνης. Δεν γνωρίζαμε τότε, δεν το γνωρίζαμε τότε αυτό, αλλά το, το σημαντικό είναι ότι αναρωτηθήκαμε πώς μπορούμε αυτό το όραμα να το, να το δοκιμάσουμε στην πράξη, τότε, εμέσω πολέμου και διαπιστώσαμε ότι γίνεται. Είναι κάτι που έγινε εφικτό και μπορέσαμε έτσι να εντοπίσουμε κάποιες πολύ βασικές αρχές. Οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι, οι πιο οι αποσπασμένοι άνθρωποι είναι αυτοί που αιτήθεται και στη βία πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη επικοινωνία μεταξύ των πολιτών και από τις δύο πλευρές του μετρόπου. Και αυτό πρέπει να γίνεται με τη συνεργασία και με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, των θεσμών, των κυβερνήσεων. Δύο φράσεις ακόμα. Ήταν επίσης σημαντικό να ρωτηθούμε όχι μόνο το τι, αλλά και το πώς. Πώς μπορούμε να ε, αποδομήσουμε αυτή την κουλτούρα του φόβου ε, και της ε, έλλειψης εμπιστοσύνης και του θυμού. Τρία-τέσσερα χρόνια μετά η δουλειά μας, την περιφέρειά μας, ήταν η πλέον επιτυχής ε, ειρηνευτική διαδικασία. Όταν η Ανατολική Κροατία μπόρεσε να επανενταχθεί στην Κροατία ε, χωρίς πόλεμο με μια ειρηνευτική διαδικασία. Και αυτό ξεκίνησε από τα κάτω. Με βάση λοιπόν αυτή την εμπειρία, πραγματικά πιστεύω ότι μπορούμε να, δώσουμε, να εμπνεύσουμε την Ευρώπη για το μέλλον, αλλά και τα Δυτικά Βαλκάνια. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε την αίσθηση, πρέπει να έχουμε μια αίσθηση σήμερα για το ποιο μέλλον θέλουμε. Ευχαριστούμε πολύ Κατερίνα Κρουχόνια. Ε, θα δώσουμε τώρα το λόγο στην δόκτωρα Κριστίνα Μπάσ, η οποία είναι Visiting Fellow από το London School of Economics. Καλό απόγευμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής ΦΑΜΕ για την οργάνωση της σημερινής ε, ακρόασης ε, και να σας πω Ε, και να σας μιλήσω για την ε, μελέτη μας όσον αφορά ε, τον ρόλο των γυναικών στις διαδικασίες ειρήνης. Να σας πω ότι γεννήθηκα σε αμερικανική στρατηγική οικογένεια και από τις δύο πλευρές ήταν στο στρατό και ο πατέρας μου είναι συνταξιούχος αξιωματικός, σε αποστρατεία τέλος πάντων. Επομένως ε, η πορεία μου ξεκίνησε με τη σκέψη πώς θα μπορούσα να συμβάλλω και να προωθήσω την ειρήνη και πώς θα μπορούσα να προωθήσω τη συμμετοχή των γυναικών σε αυτές τις διαδικασίες. Έχουμε μαζί μας σήμερα ε, ένα αντίγραφο της έκθεσης που ε, προετοιμάσαμε. Και αν θέλετε ε, μπορούμε και διμερώς μετά ε, να συζητήσουμε ορισμένα θέματα. Ε, δεν είναι πολύ ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου, γι' αυτό συγχωρέστε με εάν λόγω στενότητος χρόνου δεν μπορέσω να αναφερθώ σε όλα αυτά θα ήθελα, όσα θα ήθελα. Ε, τρία στοιχεία προκύπτουν από την έκθεση. Ε, η κατάσταση των ένοπλων σειράξεων, δεύτερον ε, το θεματολόγιο των γυναικών σε σχέση με την ειρήνη και τρίτον η συμπερίληψη των γυναικών στις διαδικασίες ειρήνευσης ε, και κυρίως στην διαδικασία στην Συρία και στη Ρουάντα. Ξέρουμε ότι έχει πολύ ε, ακολουθεί φθήνουσα πορεία ε, η ε, κατάσταση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουν γίνει πιο περίπλοκοι οι πόλεμοι. είναι πόλεμοι οι οποίοι διαρκούν και μάλιστα το διασωρινακό έγκλημα και η κλιματική αλλαγή εντείνουν πολύ συχνά την ήδη δύσκολη κατάσταση. Είναι πολλές ε, οι κρατικές σειράξεις, ε, αλλά και οι μη κρατικές έχουν, ε, ακολουθούν αυξητική τάση. Το, 2018 6,5 ε, εκατομμύρια άνθρωποι χρειάστηκε να μετακινηθούν. Σύμφωνα με την ε, Στοκχόλμη και το σχετικό Ινστιτούτο, 1,73 ε, δολάρια δόθηκαν το 2018 σαν δαπάνες πολέμου. Όσον αφορά δε, από το, τι, τι, τα, μεγάλες μετακινήσεις οπλισμών, αυτή το 18 ήταν 14,5% περισσότερο από ό,τι το 14. Η Γερμανία, η Γαλλία, ε, η Κίνα είναι ε, από τους μεγαλύτερους εξαγωγούς ε, όπλων και αντιπροσωπεύουν το 72% των εξαγωγών. Επίσης, ε, το δεύτερο στοιχείο είναι το θεματολόγιο για τις γυναίκες ε, στην 1325, ε, στο 1325 ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών αναφέρεται ότι οι γυναίκες έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν το θεματολόγιο όσον αφορά την ειρήνη. Αναφέρεται κυρίως το θεματολόγιο αυτό στην σημαντική αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στις διαδικασίες ειρήνευσης, αναφέρεται σε συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά τις γυναίκες και τα παιδιά, ε, τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα παιδιά, ε, κάνει έκκληση στα κράτη να λάβουν αποτρεπτικά μέτρα ε, και να υποστηρίξουν πολιτικές οι οποίες θα δείχνουν ευαισθησία σε σχέση με τα φύλλα. από, το, από τη στιγμή που ε, έγινε δεκτό το ψήφισμα 1325, 73 εθνικά σχέδια δράσης έχουν ε, διατυπωθεί ε, και όλα τα μέτρα αυτά καταδεικνύουν ότι η συμμετοχή των γυναικών σε ειρηνευτικές διαδικασίες μπορεί να αποτελέσουν σημαντικό όχημα για την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική πρόοδο. Ε, ωστόσο, τα εθνικά σχέδια δράσης ε, δεν ε, αναλύουν αρκετά το θέμα των στρατιωτικών δαπανών και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν στις γυναίκες και τα παιδιά, καθώς επίσης και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι δαπάνες σχετικά με τον οπλισμό, μεταφορές οπλισμού κλπ. Υπάρχουν κράτη τα οποία ζητούν την ε, μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών, αλλά σιωπηρά υποστηρίζουν την διεύρυνση της, του εμπορίου των όπλων και της μεταφοράς των ε, όπλων. Δεν ε, είναι δυνατόν να έχουν σοβαρή πολιτική. Το ίδιο ισχύει και για χώρες οι οποίες υποστηρίζουν σιωπηρά έστω την, το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας ή άλλες χώρες χώρες οι οποίες ε, έχουν εντελώς ε, ειδική αντιμετώπιση των ε, γυναικών. Βεβαίως είναι σημαντικό να πούμε ότι ένα ασφαλές περιβάλλον είναι σημαντικό για την κοινωνική ανάπτυξη ή την ανάπτυξη ελεύθερων διαδικασιών. Γι' αυτό λοιπόν μας προβληματίζει ιδιαίτερα η διεύρυνση των πολέμων ή των σειράξεων. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ε, δυνατόν να ε, ε, δεχτούμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση σύμφωνα με την οποία είναι πολύ μακρές οι ειρηνευτικές διαδικασίες με μέσο όρο την πενταετία από την έναρξη του διαλόγου μέχρι την υπογραφή των ειρηνευτικών συμφωνιών. Θα πρέπει να βρεθούν περισσότερες λύσεις ή πιο ολιστικές λύσεις. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη υπάρχει 20% αύξηση της ε, δυνατότητας επίτευξης ειρηνευτικής διαδικασίας ε, στα δύο χρόνια ε, και και πάνω από 15 χρόνια διάρκεια της ειρήνης μετά από ειρηνευτική διαδικασία εάν σε διαδικασία συμμετέχουν γυναίκες. οι γυναίκες έχουν ε, ε, ηγετικό ρόλο όσον αφορά ε, διαδικασίες παρατήρησης ή διαμεσολάβησης. Παραδοσιακά παίζουν σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες προσαρμογής της ειρήνης ή της δικαιοσύνης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις, στις ομάδες διαπραγμάτευσης να συμμετέχουν και γυναίκες έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία αυτά

και θα πρέπει να ε, συμμετέχουν γυναίκες έτσι ώστε ε, να είναι πιο σαφής η εικόνα των υποχωρήσεων που μπορούν ε, να γίνουν. Οι γυναίκες επίσης είναι σημαντικές σε διαδικασίες οι οποίες διεκδικούν είτε πρόληψη είτε ισότητα των φύλων είτε πρόσβαση στην δικαιοσύνη ή στην υγεία πολύ ε, συχνά εθνικές ε, και εθνοτικές μάλλον ε, και εθνοτικοί και θρησκευτικοί διαχωρισμοί, ε, ανισότητες και λοιπά μπορεί να αποτελέσουν το έναυσμα της βίας και κατά αυτήν την έννοια η ε, πολυμορφία και η διαφοροποίηση με συμμετοχή των γυναικών μπορεί να διευκολύνει ε, τις διαδικασίες. Η καλλιέργεια συμμετοχικού περιβάλλοντος όπου όλα τα μέλη της, και τμήματα της κοινωνίας κοινωνίας θα συμμετάσχουν ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης ε, η ιδιοκτησία όλων των διαδικασιών μπορεί να διευκολυνθεί μέσα από την παρουσία των ε, γυναικών. Επίσης είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ε, τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει οι γυναίκες ε, όταν διαδηλώνουν κατά των κυβερνήσεων ή όταν ε, συμμετέχουν σε διαδικασίες εξομάλυνσης όπως ας πούμε στην Ρουάντα ή στην Συρία οι γυναίκες εκπροσωπούν 70% του, του πληθυσμού στην ε, Ρουάντα και επομένως ήταν πάρα πολύ σημαντικές ε, στην ανοικοδόμηση και ανασύσταση της ε, χώρας το Σύνταγμα του 2003 στην Ρουάντα υπογραμμίζει ε, την συμμετοχή των γυναικών με συγκεκριμένη ποσόστοση ε, σε όλες τις ε, διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Επίσης, ε, συμμετείχαν ε, γυναίκες από όλες τις περιφέρειες και από όλα τα χωριά στην ε, διαβούλευση για, την, για, το νέο σύνταγμα. Στις εκλογές του 2003, 40% των εδρών κερδίθηκαν από γυναίκες. Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι η προώθηση των γυναικών σε κρίσιμα πεδία ε, έχει αντιστρέψει παραδοσιακές διαδικασίες ε, στην ε, Ρουάντα, γιατί η συμμετοχή γυναικών σε διαπολιτισμικές ή πολιτικές διαδικασίες είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Το 2011 ξεκίνησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις Εκεί ε, είχαμε ε, ε, χρήση το, είχαμε βολές κατά των, κατά των αμάχων, καθώς επίσης και μαζική χρήση των συλλήψεων και των βασανισμών οι γυναίκες ε, και τα παιδιά ε, είναι ε, αυτές οι οποίες αναγκάστηκαν ακριβώς λόγω του ότι οι άντρες είτε εξαφανίστηκαν είτε φυλακίστηκαν είτε και έχασαν τη ζωή τους, αναγκάστηκαν λέω να αναλάβουν τα ενία της οικογένειας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση των οικογενειακών δικτύων και των, των οικονομικών καταστάσεων, αλλά οδήγησε και σε ε, μια νέα μορφή εκμετάλλευσης ε, ε, και όσον αφορά τους μισθούς και όσον αφορά τις διαδικασίες, εργασίας και τις εργασιακές συνθήκες. Επομένως δεν ολοκληρώθηκαν κατά κάποιο τρόπο οι προσδοκίες των γυναικών. Η Συμβουλευτική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών που ανέλαβε την διαδικασία ε, ειρήνευσης ε, ε, προσπάθησε να βρει λύσεις σε όλα τα ζητήματα τα οποία ανέφερα μέχρι τώρα. Σε τοπικό επίπεδο επίπεδο ε, και παρά την, ε, τον κίνδυνο ε, σύλληψης ή απαγωγής από φιλοκυβερνητικές δυνάμεις έγιναν πολλές προσπάθειες για να μοιραστούν φάρμακα, για ενημέρωση κλπ. Τώρα, η συμφιλίωση και η δικαιοσύνη μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον ε, συνεχών ε, ε, παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πώς μπορεί να κερδιθεί μακροπρόθεσμα μέσα από την συμμετοχή των γυναικών και την συμπερίληψη των γυναικών σε μια πιο συμπεριληπτική και χωρίς βία κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Κριστίνα Μπέιτς. Και τώρα θα δώσω τον λόγο ε, στη, στη Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Ένα σημείο που είναι καινούριο είναι αυτά που είπατε για την Δυτική Σαχάρα. Γιατί μιλήσαμε για την εμπορική συμφωνία με τη Δυτική Σαχάρα και με το Μαρόκο και δώσαμε την έγκρισή μα για αυτή τη συμφωνία, παρόλο που δεν υπάρχει συμμετοχή των ατόμων στην Δυτική Σαχάρα ή επαρκής συμμετοχή ούτε των ανθρώπων ούτε των γυναικών. Η ερώτησή μου είναι που απευθύνεται σε εσά και συγκεκριμένα στην ε, ομιλήτρια που έκανε αναφορά στην ε, Δυτική Σαχάρα. Αυτή η συμμετοχή στις ειρηνευτικές διαδικασίες στα θέματα εμπορικών συμφωνιών σε, περίοδους η συμμετοχη στι ειρηνευτικε διαδικασίε στα θεματα εμπορικων συμφωνιων σε περιοδους ειρηνης θα μπορούσαν να υπάρξουν ε, κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης για να μπορεί να υπάρξει συμμετοχή, γιατί κατάλαβα και αρκετά επώδυνα ότι όταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνουμε λόγο για το εμπόριο, δεν ε, λάβαμε υπόψη τους πολίτες, τις γυναίκες στη Δυτική Σαχάρα και πώς μπορούμε να πετούμε τη συμμετοχή του σε ε, ερευνητικέ διαδικασίε όταν δεν συμμετέχουν σε άλλε διαδικασίε που άπτονται τη καθημερινή του ζωή, όπω είναι το εμπόριο. Θεωρείτε ότι είναι, κάτι, είναι, κάτι, είναι δύο τελείω διαφορετικά θέματα, γιατί δεν ε, είναι κάτι αυτό που σα είπα που ταιριάζει στη δικασία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Στην κυρία Μπαρζάνου λόγος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί καλεσμένοι, θέλω να σας ευχαριστήσω που μοιραστήκατε μαζί μας τη γνώση σας. Θα ήθελα να σας πω ότι όλα όσα άκουσα σήμερα είναι συγκινητικά. Σας νιώθω πραγματικά γιατί κατάγομαι από μια περιοχή της ε, Ευρώπης που βρισκόταν σε πόλεμη κατάσταση πρόσφατα. Πολλά από αυτά που άκουσα εδώ σήμερα τα έχω αισθανθεί στο πετσί μου. Γι' αυτό ε, με αγγίζει πολύ συναισθηματικά αυτή η συζήτηση. Έχουν περάσει 20 χρόνια από τον πόλεμο και πάντα κάνουμε αναφορά στην αλήθεια και στη δικαιοσύνη ως κίνητρα, γιατί πολλά θύματα δεν βρήκαν το δίκιο τους ούτε την αλήθεια. Έχω υπάρξει εισηγήτρια του Κοινοβουλίου για το ψήφισμα για τα Δυτικά Βαλκάνια. Η Επιτροπή ενέκρινε εδώ και λίγο καιρό το ψήφισμα όμως ακόμα δεν έχει τεθεί στην ε, μερίσια διάταξη της Ολομέλειας. Ανησυχώ ότι ενδεχομένω να μην περάσει το ψήφισμα στη διάρκεια αυτής της θητείας και αυτό θα ήταν πραγματικά κρίμα γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες χώρες που ενδεχομένως να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ένταξης ή προένταξης και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις χώρες αυτές και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τις βοηθήσουμε γιατί οι πολίτες τους έχουν ζήσει πολέμους, έχουν υποστεί τις συνέπειες των πολέμων και ακόμα και σήμερα θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, να τους βοηθήσουμε να οργανώσουν τις κοινωνίες τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να μπορέσουν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σας πω και άλλα, δοθείς της ευκαιρίας, ε, για την έκθεση γιατί είχε κυρίως να κάνει με τις ε, χώρες σε μεταπολεμική περίοδο και πώς ε, είναι η κατάσταση τη γυναίκε σε αυτέ τι χώρε. Είναι γενική, κάνει λόγο για σταθεροποίηση, διαδικασία σταθεροποίηση, διαχείριση κρίσεων, το ρόλο των γυναικών και την εφαρμογή ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για την, ε, του Συμβουλίου Ασφαλής για την ε, ασφάλεια των γυναικών. Δίνεται επίσης έμφαση στη συμμετοχή των γυναικών στην ε, λήψη αποφάσεων. Και τι εννοούμε με αυτό, ότι οι γυναίκες θα πρέπει να συμμετέχουν και να εκπροσωπούνται σε τοπικά συμβούλια, τοπικά κοινοβούλια όπου λαμβάνονται αποφάσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που αφορούν κυρίως ε, τις γυναίκες σε χώρες που έχουν πληγεί από πόλεμο, όπου οι καταστάσεις είναι δυσχερείς, γυναικες θύματα πολέμου, βιασμών κτλ. Αυτές οι καταστασεις ειναι δυσχερεις γυναικέστήματα θυματα πολεμου βιασμων κτλ αυτες οι γυναικες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην διαδικασία λήψη αποφάσεων και να μην βλέπουμε μόνο άντρε να λαμβάνουν αποφάσεις εκ μέρους τους. Από την άλλη όμως δεν θέλουμε κάποια θέματα να γίνουν αποκλειστικά θέματα γυναικών. Είναι σημαντικό οι γυναίκες θύματα να έχουν πρόσβαση επίσης στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιστάσεις για τις οποίες κάνουμε λόγο στην Επιτροπή στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, όπου οι γυναίκες δεν έχουν τους μηχανισμούς, τους τρόπους για να βελτιώσουν τη θέση τους θύματα πολέμου και περισσότερο θύματα βιασμών. Αυτές οι γυναίκες στιγματίζονται και δεν ε, έχει γίνει κάτι ως προς αυτό. Θα πρέπει να υπάρξει μία νομοθετική διάταξη που να αφορά, για τις, ε, αφορά τις γυναίκες θύματα πολέμου. Γιατί αλλιώ ο κάθε δικαστή μπορεί να δώσει τη δική του ερμηνεία. Θέλουμε μια συγκεκριμένη επομένω νομοθετική ε, διάταξη για τι γυναίκε θύματα πολέμου στη Σερβία. Ο διάλογο μεταξύ Βοσνίας, Ζεγοβίνης και Σερβίας προωθείται, προάγεται, γιατί υπάρχει μια πολιτική σύγκρουση ακόμα ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες. Θα θέλαμε να εμπλακούν και σε αυτή τη δικασία οι γυναίκες. Όσον αφορά τη Μακεδονία και το Μοντανέγκρο, το Μαυροβούνιο, δεν έχουμε επαρκή αριθμό μη κυβερνητικών οργανώσεων που να συμπεριλαμβάνονται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Σε όλες τις χώρες της Βαλκανικής υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό κάτι που θα πρέπει να καταγγείλουμε γιατί δεν είναι μόνο οι τοπικές οργανώσεις που θα πρέπει να αναλάβουν αποκλειστικά αυτά τα θέματα σε <clears throat> χώρες μετά τον πόλεμο. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτή τη διαδικασία. Επίση, δόθηκε έμφαση και στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στι χώρε των Δυτικών ε, Βαλκανίων. Βλέπουμε έναν ηθικό διχασμό, εθνοτικό μάλλον διχασμό στα, σχολείο, στα σχολεία. Και αυτό εμποδίζει την ειρηνευτική διαδικασία. Όταν διασπείρουμε προκαταλήψεις, τότε είναι δύσκολο να στήσουμε τα παιδιά για την ειρήνη και τη συνύπαρξη. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη σημασία της εκπαίδευσης που είναι το μέσο της πρόοδου σε αυτές τις χώρες. Η Κροατία, από την οποία κατάγομαι, δεν είναι κομμάτι των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά η Κροατία έχει παρόμοια θέματα με τις χώρες αυτής της περιοχής. Όπως είπα και στην αρχή, η Κροατία χτυπήθηκε από τον πόλεμο και ακόμα προσπαθούμε για την οικοδόμηση ειρήνης. Υπάρχουν πολλοί, πολλοί άρθιμοι πολίτες στην ε, Κροατία που δεν έχουν βρει τα αγαπημένα τους πρόσωπα, που δεν έχουν βρει το δίκιο τους και που ακόμα περιμένουν ε, δικαστικές αποφάσεις. Δεν είναι ικανοποιητική καθόλου η κατάσταση. Θα ήθελα να κάνω έκκληση στον συντονιστή του ΕΛΚ και σε όλους τους άλλους να εγκρίνουν την έκθεση μέχρι το λήξη αυτή της θητείας, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τις κυβερνήσεις τους να πράξουν τα ανάλογα και μερικώς να επιλύσουν τα θέματα τα οποία έφτιαξα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τώρα την Julie Ward παρακαλώ. Δύο-τρία λεπτά όμως, ε, όχι παραπάνω, γιατί θέλω να δώσω το λόγο ξανά και στους εμπειρογνώμονες για να απαντήσουν. Παρακαλώ κυρία Ward. Θα είμαι σύντομη, αν και έχω πολλά να πω. Πρώτα απ' όλα πραγματικά εκτιμώ ότι λαμβάνει η χώρα αυτή η ακρόαση σήμερα και ζητώ συγγνώμη για την πολύ έτσι συχνή συμμετοχή. Χαίρομαι που η μόνη οι ευρωβουλευτέ που μένουν εδώ πέρα είναι από τη δική μου πολιτική ομάδα, του Δημοκράτε. Ε, είμαστε εξαιρετικά θετικοί στο έργο που κάνουμε ε, για τα δικαιώματα των γυναικών, ε, για την ενδυνάμωσή του. Μόνο σε δημοκράτε νομίζω είναι εδώ. Έτσι πρέπει να το πούμε και αυτό. Σε ό,τι αφορά την Λίγα της Ειρήνης και της ε, Ελευθερίας των Γυναικών Έχω πολλούς φίλους εκεί και μου λένε ότι φτάνουν πολλές νέες γυναίκες στην οργάνωση αυτή και ότι πραγματικά μεταλλάσσεται ε, η οργάνωση αυτή και ό,τι αφορά τη συμμετοχή της ε, και την παρουσία της στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Να μας, δώσετε, να μας πείτε λοιπόν κάτι περισσότερο για τις νέες γυναίκες. Θέλω να μιλήσω γι' αυτό, επειδή είπατε όλοι πολλά σημαντικά ζητήματα ε, για το δημογραφικό θέμα ε, και έχουμε στο πάνελ, τι έχουμε τελικά όμως, λευκές γυναίκες, με μεσαία τάξη, έτσι. Ούτε τόσο νέοι, ε, τόσο νέες γυναίκες, ούτε από άλλα, ε, από άλλα κοινωνικά στρώματα. Θα ήταν καλύτερο λοιπόν να υπάρχει μια εκπροσώπηση αυτών που, για τους οποίους... Ε, ζητάτε δικαιώματα. Εγώ ασχολούμαι με τις σχέσεις με τη Βοσνία και την ε, τη Βοσνία Τσογοβίνη και το Κοσφοπέδιο, συνήθω αυτοί που ε, διαχειρίζονται την ειρήνη είναι αυτοί που έκαναν και τον πόλεμο. Οι άντρε δεν αφήνουν εύκολα την εξουσία, στι διαθέσει βρίσκονται, αυτοί είναι που έχουν τον έλεγχο, θέλουν πάντα να είναι από πάνω και είναι δύσκολο να πιστούν άντρε οι οποίοι πάντα είχαν την εξουσία να την δώσουν. Αυτό ισχύει και για εμά, του αριστερές και δημοκράτε ε, και στην πολιτική μα ομάδα και στη δική μα πολιτική οικογένεια. Ε, είναι κάτι το οποίο, ε, για το οποίο δίνουμε μια μάχη, μια σκληρή μάχη για να συμβεί κάτι τέτοιο. Γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποιε χώρε ίσω η Άννα να πει τώρα γι' αυτό, υπάρχει ένα μοντέλο πάντως φεμινιστικής εξωτερικής πολιτικής που υπάρχει στη Σουηδία και θέλω να πω τιμής Έχω συναντήσει πολλές ε, ε, Σουηδέζες πολιτικούς ε, που πραγματικά αυτή τη στιγμή δείχνουν το δρόμο και κάνουν αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε όλοι. Να υπάρχει μια φεμινιστική εξωτερική πολιτική. Και αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα είχαμε πολύ περισσότερες γυναίκες σε αυτές τις θέσεις και πολύ λιγότερους πολέμους. Πραγματικά με ενδιαφέρει το case study σας για τη Συρία. αναφερθήκατε στον ρόλο του YPJ, αλλά λέτε απλώς ότι είναι μαχητές. Δεν λέτε για την, την ε, εμπειρία, το, το πείραμα της Ροζάβα, όπου οι γυναίκες είναι αυτές που οικοδομούν την κοινωνία ε, σε αυτήν την περιφέρεια. Ε, αυτή, το, αυτό το πείραμα το δημοκρατικό δείχνει ότι όταν οι γυναίκες αναλαμβάνουν τα πράγματα έχουμε διαφορετική κοινωνία ακόμα και σε εποχή πολέμου αν η κοινωνία. Ε, και πραγματικά ε, στενοχωρέθηκα που δεν το είπατε. Εγώ έχω πάει εκεί. Ε, τον περασμένο Μάιο ήμουν στη Ρουζάβα στην, σε μια αντιπροσωπεία γυναικών για την ειρήνη. Πείτε τα αυτά στην έκθεση. Μην μιλάτε μόνο για γυναίκε ω θύματα ή, ή ως μαχητές. Πείτε τι γίνεται στη Ρουζάβα. Γιατί είναι μια πραγματικά εξαιρε... ένα εκπληκτικό ε, παράδειγμα. Η Λέιλε δεν είναι εδώ, η Λέιλε δεν είναι εδώ σήμερα επειδή έκανε απεργία διότι ο αγώνα των Κούρδων συνεχίζεται, διότι οι άνθρωποι που θέλουν διαφορετικού, μια διαφορετική κοινωνία όπω οι Κούρδοι, ένα περιβαλλοντικό μοντέλο που βασίζεται στην ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, έχουν μείνει εκτό διαδικασία. Ε, και όλα αυτά βεβαίω ε, σχετίζονται και με τις τουρκικέ εκλογές το Σαββατοκύριακο. Αυτό που είπε η Μπιλιάν είναι πολύ σημαντικό, διότι αναφέρθηκε στην εκπαίδευση. Όσοι από εμά συμμετέχουν στην Επιτροπή για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό γνωρίζουμε ότι χρειάζεται πλέον ηθαγένεια ε, ευρωπαϊκή, χρειάζεται εκπαίδευση για την ισότητα των δύο φύλων, για την ειρήνη. Πρέπει να μιλάμε για αυτά τα πράγματα ήδη στα σχολεία, τα, στα, παιδιά από τα σχολεία. Ε, το πρόγραμμα Erasmus Plus, παραδείγματο χάρη, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλου μα να ενισχύσουμε ε, τις ιδέες που έχουν για την Ευρώπη οι νέοι για να καταλάβουν ότι η Ευρώπη είναι ένα ειρηνικό σχέδιο και ότι όλοι έχουμε ευθύνη γι' αυτό ε, να μιλήσουμε τότε δηλαδή για την ειρήνη. Τώρα, εν ώψη της επόμενης ε, όταν θα έχουμε τον, τον κοινό χώρο εκπαίδευσης, τον ευρωπαϊκό, θα είναι η στιγμή και για τις γυναίκες να πούν ότι θέλουμε η Ευρώπη να είναι ειρηνικό σχέδιο και ο ρόλος των γυναικών σε αυτό το σχέδιο πρέπει να ενισχυθεί. Αναρωτιέμαι πόσοι από εσά γνωρίζετε ε, το Brussels Peace Pledge, η έκκληση για την ειρήνη των Βρυξελών. Ε, εγώ το 2014 ήρθα εδώ και κανείς δεν μου είπε ότι οι βουλευτές είχαν ε, υπογράψει εδώ στο Κοινοβούλιο αυτή την έκκληση. Ε, και υπάρχουν ακτιβιστές από τη δική μου περιφέρεια που προσπαθούν να αναζωογονήσουν ενδιαφέρον για αυτό. Ε, νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει, είναι κάτι πρακτικό έτσι ώστε να ε, έτσι οι ακτιβιστές σε τοπικό επίπεδο να μπορέσουν να συνδεθούν με τους επόμενους ευρωβουλευτές της επόμενης θητείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Ward. Και τώρα απευθύνομαι σε όλα τα μέλη ε, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εάν όχι, να δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονές μας. Να ακούσουμε τα σχόλιά σας ή τις αντιδράσεις σας. Παρακαλώ. Η κυρία Μαγκαγιών, ε, δύο-τρία λεπτά ο καθένας παρακαλώ, διότι έχουμε λίγο χρόνο ακόμα για την ακρόαση αυτή. Ναι, θα είμαι σύντομη στα ισπανικά. Ευχαριστώ για το ερώτημα για την ε, Δυτική Σαχάρα. Είναι ένας από τους ξεχασμένους πολέμους. Από το 1975 άνθρωποι που ζουν στους καταβλισμούς του Τιντούφ και κάποιοι άλλοι που ζουν σε μια χώρα που δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματά τους, τα δικαιώματά τους για την αυτοδιάθεση, διότι τα, ε, η Δυτική Σαχάρα έχει δικαίωμα αυτοδιάθεσης, είναι ένα έδαφος ε, το οποίο είναι απικία. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι ότι μια ομάδα γυναικών από τη Δυτική Σαχάρα, νέων γυναικών βεβαίως και αυτό είναι παράγοντας διάκρισης έτσι, να συμμετέχουν οι γυναίκες, ε, οι νέες, αλλά μην μας πετάτε έξω εμάς τις πιο ηλικιωμένε. έτσι. Λοιπόν, αυτή η ομάδα των γυναικών από τη Δυτική Σαχάρα που που σπουδάζουν στην Ισπανία γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση και από τις δύο πλευρές του τείχου και θέλουν να παρέμβουν στις συζητήσεις, θέλουν να έχουν το δικαίωμα να παρέμβουν με βάση και τις, ψηφίσματα των Εθνών θεωρούν ότι μπορούν να συνεισφέρουν να δώσουν μια νέα προσέγγιση ό,τι αφορά αυτή τη σύραξη. Είναι περίπλοκη αυτή η σύραξη. Βεβαίω υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. το πετρέλαιο, η παραγωγή, ε, που μπορεί να προσφέρει η Δυτική Σαχάρα. Υπάρχουν τα σφαίροντα της Γαλλίας, του Μαρόκου, της Ισπανίας, της Αλγερίας. Εμπλέκονται και ζητήματα τρομοκρατίας. Στις με το Μαρόκο. Όμως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ομάδες νέων από τη Δυτική Σαχάρα που δεν βλέπουν παρόν, δεν βλέπουν μέλλον και σκέφτονται να ξαναπάρουν τα όπλα. Ε, και η ελπίδα αυτών των γυναικών είναι να τύχουν υποστήριξη ως ομάδα και να μπορέσουν να συμμετάσχουν και σε ανταλλαγή, ανταλλαγές με άλλες γυναίκες από το Μαρόκο, να μπορέσουν να συνεργαστούν. Εδώ για, για πολύ καιρό θεωρήθηκε ότι οι γυναίκες της Δυτικής Σαχάρας ήταν οι πιο προ, του αραβικού κόσμου, όμως αυτέ οι νέες γυναίκες λένε ότι και ε, εκ νέου ε, υποβάλλονται σε ένα καθεστώς ε, φιλής όταν ε, επιστρέφουν στις οικογένειάς τους ουσιαστικά ε, είναι υποταγμένες και μπαίνουν σε μια ε, κατάσταση όπου δεν αναγνωρίζεται καν ανήλικη, το του ανήλικου ε, βεβαίως ταυτόχρονα υπερασπίζεται την αυτοδιάθεση πρέπει λοιπόν να, να πιστεί το μέτωπο πολυσάριο ότι δεν είναι κατά της αυτοδιάθεσης θέλουν να προσθέσουν και τα προβλήματα των γυναικών όμως. Τα δικαιώματα των γυναικών στην υπόθεση αυτού του δικαίωμα να έχει κάποιος ε, μία ε, εργασία, να μπορεί να μπει και να βγει από το έδαφος και να μην υπόκειται στον νόμο της Σαρία που επιβάλλεται στη Δυτική, στη Σαχάρα σιγά σιγά. Όλο και πιο συχνά λοιπόν έρχονται και νέες γυναίκες στη Λίγα μας. Είναι όμως μια οργάνωση που υπάρχει εδώ και 100 χρόνια. Ε, στην Αφρική πάντως υπάρχουν πολλές ομάδες γυναικών πολλά τμήματα εθνικά. Η Τζο Ιόνισον, η, η πρόεδρος μας, είναι από την Ιγυρία. Πιο νέοι άνθρωποι και εμείς ευχαρίστως τους υποδεχόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δύο σύντομα σχόλια. Το πρώτο πιο γενικό ε, σχετικά με την ερώτηση όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες με τη Δυτική Σαχάρα. Ε, η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης οπωσδήποτε θα πρέπει να υπόκειται ε, σε ενδελεχή ανάλυση όλων των στοιχείων των χωρών, καθώς επίσης και ανάλυση των συνθήκων σύραξης, καθώς επίσης και συμμετοχή Όλη τη κοινωνία και όχι μονάχα της αστικής ε, κοινωνία. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται ε, ε, έμφυλη ανάλυση έτσι ώστε σε οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία ή οποιαδήποτε άλλη μορφή παρέμβασης να υπάρχει και αυτό το ε, στοιχείο ε, και μονάχα ε, εάν μπορεί να, εάν δεν γίνει τέτοια ανάλυση σύραξης δεν είναι δυνατόν να μην είναι δυνατόν να προχωράει οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση ή υποστήριξη. Επίσης πρέπει να πω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της συμμετοχής. Αν θέλουμε να έρθουν μεσολαβητές γυναίκες στις ε, ε, Βρυξέλλες. Ε, θα πρέπει να διευκολύνουμε και την συμμετοχή. Εμείς επί σειρά μηνών προσπαθούσαμε να πάρουμε βίζα για κάποιες γυναίκες για να έρθουν στις Βρυξέλλες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει κανείς τέτοιου είδους άδειες ταξιδιού κτλ θα πρέπει, ε, θα πρέπει, και ε, ε, θα πρέπει όλοι να βοηθήσουν γιατί όλα αυτά σημαίνουν χρήματα, σημαίνουν διαδικασίες θα πρέπει οπωσδήποτε νωρίς ε, να αποφασίζετε ποιες γυναίκες θέλετε να καλέσετε. Εάν θέλετε να έρθουν αυτές οι γυναίκες, αν, θέλουν, αν θέλουμε να τις βγάλουμε από τη σκιά που τις βαραίνει, θα πρέπει να τις βοηθήσουμε, αλλά θα πρέπει έγκαιρα να ξεκινήσουμε. Η κυρία Ποητάνεν, ευχαριστώ πολύ και εγώ ε, θα πω δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα θα συμφωνήσω με αυτά που είπε η Λόρα όσον αφορά την πρόκληση της ε, αντιπροσώπευσης. Ε, βεβαίως εμείς είμαστε πάντα στην ε, διάθεση όλων των γυναικών που δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά μέσα σε πολύ σκληρές πραγματικότητες ο τρόπος που βλέπουμε τις ε, γυναίκες ε, στις ε, διαδικασίες ειρήνευσης είναι πάρα πολύ σημαντικός και είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται ο ρόλος τους ως στη διαδικασία οικοδόμησης ε, ειρήνης αλλά και διατήρησης της ειρήνης. Δεν ξέρουμε πολύ καλά ε, την κατάσταση και μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι αν ε, βάλουμε πολλές γυναίκες μαζί θα έχουν όλες ε, την ίδια άποψη όμως είναι μια ιδέα που θα πρέπει να σπάσει θα πρέπει να δούμε τις γυναίκες ως πολιτικά όντα και ως πολιτικούς πρωταγωνιστές και δεύτερον πολύ σύντομα η σημασία των μακροπρόθεσμων και μακρόθωρων ε, διαδικασιών όπως είναι ας πούμε η ε, εκπαίδευση. Ε, αυτά όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και εμείς τα προωθούμε. Τέλος αυτό που είπε η Λόρα, τις ευκαιρίες να, οι ευκαιρίες που πρέπει να δίνουμε στις ε, γυναίκες αυτές να μιλήσουμε για τις αξίες ε, που είναι παγκόσμιες αξίες. Ε. Νομίζω ότι όλοι είμαστε στη διάθεσή σας για να δουλέψουμε όλοι μαζί, για να τα προωθήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κρούχωνια. θα ήθελα να συνεχίσω ε, ε, ε, για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα της εκπαίδευσης για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε την ειρήνη ή να οικοδομήσουμε τον πολιτισμό, την κουλτούρα της ειρήνης χρειάζεται ε, εκπαίδευση. Εκπαίδευση για την ε, αποτροπή της βίας. Ε, επίσης, για να γίνει η εκπαίδευση στην, κατά της βίας εύκολα προσβάσιμη για τους καθηγητές, για το διδακτικό προσωπικό, για τις γυναίκες, για τα παιδιά. Στην Ευρώπη, αλλά κυρίως ε, στα Δυτικά Βαλκάνια, κάτι τέτοιο είναι απολύτως απαραίτητο. Και ένας άλλος τρόπος ε, για να ενδυναμωθεί ε, το κοινό έτσι ώστε να χτίσει ισχυρές σχέσεις είναι οι διασυνοριακές συναντήσεις ανθρώπων. Αυτό το ε, ε, πρόγραμμα κινητικότητας του έρασμου είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, σε μια περιοχή δηλαδή που δεν συμμετέχει στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να δοθούν δυνατότητες συνεργασίας, συνάντησης, ανταλλαγής απόψεων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αν γίνεται και μεταξύ των γυναικών ακόμα καλύτερα. Με τον τρόπο αυτό ε, θα συναντηθούν, θα ανταλλάξουν απόψη οι γυναίκες, αλλά και αυτές οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν και μια οικονομική υποστήριξη. Γιατί θα πρέπει να μάθουν οι μεν την εικόνα των δε. Δύο λόγια για τον πόλεμο στη Συρία. Ναι, ε, είναι ε, γεγονός ότι υπάρχουν ε, ε, γυναικείες μονάδες σε, από όλες τις πλευρές και η ίδια η κυβέρνηση στις κυβερνητικές ομάδες έχει μία ομάδα γυναικών μαχητών. Είναι γεγονός πάντως ότι ο μη ε, στρατιωτικός, μη πολεμικός ρόλος των γυναικών στη Συρία δεν έχει καταδειχθεί αρκετά. Ίσως εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε και στην χρηματοδότηση από πλευράς ε, των ε, χωρών της ε, Δυτικής Ευρώπης υπάρχουν οργανώσεις όπως το CVE που δίνουν την δυνατότητα ελέγχου των οικονομικών έτσι ώστε πραγματικά να υποστηρίζονται μονάχα ειρηνευτικές διαδικασίες. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις συμμετέχουσες ε, στο, στη σημερινή ακρόαση, να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονες, αλλά και τα μέλη της δικής μας ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Σήμερα είχαμε για μία ακόμα φορά ε, την ε, ευκαιρία να δούμε πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν γυναίκες στις διαδικασίες ε, ειρήνευσης και οικοδόμησης της ειρήνης. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει οπωσδήποτε να αντικατοπτρίζουν τα όσα συζητήθηκαν σήμερα. Είναι ανάγκη ε, να εγκρίνουμε τις σωστές αποφάσεις και όπως είπε και η Λιάννα Μπορζάν ε, θα χάσουμε εάν δεν μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτές τις αποφάσεις ε, και θα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι τον Απρίλιο στην τελευταία ολομέλεια στην ημερήσια διάταξη ότι θα συμπεριληφθεί το θέμα αυτό των Δυτικών Βαλκανίων. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία και στο μέλλον να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. με Θα συνεχίσουμε λοιπόν την συνεδρίασή μας, λέει η Πρόεδρος. Παρακαλώ πολύ καθίστε. Λοιπόν, έχουμε το σημείο 5 της ημερησίας διατάξεως ε, σχετικά με την Λέιλα Γκιούβεν Θα θυμάστε ίσως ότι στην αρχή της συνεδρίασης είπα ότι έχει πολύ σημαντικά προβλήματα υγείας γιατί ε, έχει απεργία πείνας εδώ και κάποιους μήνες και δεν είναι σε θέση να ε, είναι εδώ. Θα την αντικαταστήσει η κυρία Σερμάλ Καμίλ Μπέι, η οποία θα μας ε, δώσει, θα, θα μας μιλήσει εκ μέρους της. Türkiye'den geliyorum. İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay. Hi dear friends. I would like... Αγαπητοί φίλοι, τους επαναστατικούς μου χαιρετισμού, το όνομά μου είναι Κεμάλ E, Από τη Σμύρνη. Είμαι. Yaşadık ve ben onun havasıyla, rüzgarıyla burada geliyorum, buraya geldim. Thank you very much for... Σας ευχαριστώ πολύ. Πώς επιτροπή μας καλέσατε σήμερα εδώ. Πρόσφατα είχαμε τοπικές εκλογές στην Τουρκία και είμαι εδώ έχοντας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 αυξάνεται η φθαρχικότητα. Φθαρχικά ε, καθόλου σε όλο τον κόσμο, το ισχύει και στην ε, Τουρκία. Αγωνιζόμαστε ενάντια σε αυτό το κατεστημένο και σηκώνουμε το αναστημά μας, υψώνουμε το αναστημά μας. Ε, bu konuda The most for in Turkey. Το πιο σημαντικό για εμάς στην Τουρκία είναι τα θέματα των γυναικών και το κουρδικό ζήτημα που δυστυχώς δεν έχει επιληθεί γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά στον τομέα της δημοκρατίας και σε όλα τα υπόλοιπα στην Τουρκία. En önde de Leyla Güven, Hakkari milletvekilimiz duruyor. Women are leading for the struggle. Ηγούνται του αγώνα αυτό οι γυναίκες και η Λέλα είναι, το προ... είναι η πρωτεργάτης αυτής της προσπάθειας. Pratik çözümün yaşanabilmesi için tecritin kaldırılması, Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması önem kazanıyor. Για να πετύχουμε την ειρήνη στην Τουρκία πρέπει να ε, σταματήσει η απομόνωση του Αμπτουλάχο Τσαλάν. Είναι ένα πολύ βασικό σημείο στο κουρδικό ζήτημα. 6 gündür ε, açlık grevinde 109 gündür e, tutsaklar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 το στις 46η μέρα της απεργίας πείνας και πολλοί άλλοι φυλακισμένοι βρίσκονται σε απεργία πείνας και ενδεχομένως το έχετε ακούσει πάρα πολλοί βρίσκονται σε απεργία πείνας σε ολόκληρο τον κόσμο όπως και στην Ευρώπη. Ε, Λέιλα ε, bu özellikle hapishanelerden tabu çıkmasını istemiyor ve Türkiye'deki bu hukuksuzluğun bitmesini istiyor. O nedenle sizlere bir mektup gönderdi. Leyla doesn't want any coffins to come out from the prisons. Η Λέιλα δεν θέλει να βγουν φέρετρα από τις φυλακές και γι' αυτό σας στέλνει αυτή την επιστολή. Şimdi okuyacak hepinizin dinlemesini talep ediyorum. Leyla Güven'in en sıcak duygularla sizleri kucaklıyor, selamlıyor. Ben de bunu buradan size iletmek istiyorum. And um, Leyla warmly hug you send. Σα στέλνει τα χαιρετίσματά τη, τα θερμά και την αγάπη τη σε όλε τι γυναίκε του Ευρωκοινοβουλίου. Και τώρα θα σα διαβάσουμε την επιστολή τη. Αγαπητές γυναίκες, όπως γνωρίζετε, εγώ και χιλιάδες άλλοι βρισκόμαστε σε απεργία πείνας. Ίσως είναι δύσκολο να καταλάβετε γιατί ενεργούμε έτσι. Μπορεί κανείς να υψώσει τη φωνή του με άλλο τρόπο. Γιατί να βλάψει τον εαυτό του. Ίσως το ρωτήσετε αυτό. Αλλά να είστε σίγουροι ότι προσπαθήσαμε πολύ σκληρά ενάντια στην απομόνωση του κύριου Τσάρλαν, Κανεί όμω δεν μα άκουσε δυστυχώ. Στην χώρα στην οποία ζούμε δεν υπάρχει ελευθερία έκφραση, ούτε καν φυσικά η ελευθερία τη ε, διαμαρτυρία. Γι' αυτό το λόγο πολλοί πολιτικοί, Κούρδοι ε, ε, πολιτικοί, διανοούμενοι, συγγραφείς και δημοσιογράφοι είναι στη φυλακή. Δικαζόμαστε για κομικοτραγικούς λόγους, όπως το να ζητάμε το τέλος της απομόνωσης στη φυλάκηση, εξαιτία του Γιώργου του λέμε του λέξη Κουρδιστάν και που υποστηρίζουμε την αυτονομία. Και γι' αυτό το λόγο πολλοί από εμά ε, βρισκόμαστε πίσω από τα σύνδερα τη φυλακή ή στην εξορία. Ω δημοκρατικά εκλεγμένη εκπρόσωπος δεν μπορούσα να βρω άλλο τρόπο πέρα από την απεργία πείνα. Θεωρώ ότι στον 21ο αιώνα οι βουλευτέ, οι πολιτικοί, οι γυναίκε και οι νέοι κάνουν απεργία πίνης για να τους ε, ακούσει η διεθνής κοινότητα. Και εγώ και οι φίλοι μου αγαπούμε τη ζωή, αλλά μια ελεύθερη ζωή και μια ισότιμη ζωή. Άκουσα ότι θα είχατε αυτή τη συνεδρίαση. Σας χαιρετίζω σε αυτή τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Θα ήθελα να βρίσκομαι εκεί για να σας απευθύνω το λόγο, αλλά η επειδή είναι στις υγείας μου δεν μου το επέτρεψε αυτό. Το ηθικό μου είναι υψηλό, αλλά δεν μπορώ να ε, αυτοεξυπηρετώ και χρειάζομαι τη βοήθεια της κόρης μου και των φίλων μου. Όταν ξεκίνησα την ε, απεργία πείνας, ήξερα το φασιστικό κόμμα δεν θα ε, άλλαζε τη στάση του. Γι' αυτό το λόγο ετοίμασα τον εαυτό μου για το αποτέλεσμα. Όπως ο Μπόμπι Σάντς, όταν ήταν στην ε, φυλακή. Έτσι και εγώ θα έδινα τη ζωή μου για τα δικαιώματα των συμπολιτών μου. Είναι η 146η μέρα της απεργίας μου και τώρα ακούτε τη φωνή μου. Γυναίκες από όλο τον κόσμο έχουν ε, δείξει την αλληλεγγύη τους, η οποία ήταν πολύ σημαντική και που μου έδωσε πολύ δύναμη. Ωστόσο, για να μείνω στη ζωή και εγώ και οι χιλιάδες φίλοι μου χρειαζόμαστε μια πιο ισχυρή φωνή. Καθώς οι νόμιμες απαιτήσει μας δεν ικανοποιούνται, φέρετρα βγαίνουν από τις, φυλακές, από τις φυλακές και οι σύντροφοί μας θυσιάζουν τις ζωές τους για να τονίσουν την απανθρωπιά και για να μας κρατήσουν ζωντανούς. Η Αγία μου έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο και η δικιά μου και των ε, συντρόφων μου. Καθώς υπάρχει ε, περιφρόνηση πραγματικά από την κυβέρνηση, από το κυβερνό κόμμα των διεθνών συμφωνιών, Αυτό αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τι γυναίκε μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν ειρηνικό κόσμο. όπου θα εφαρμόζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ισότιμα για όλους. Μπορούμε να κρατήσουμε τη σημαία που μας παραδόθηκε από τις κλάρες της, από τις κλάρες της ρόζες και τις ακίνες του κόσμου. Θεωρώ ότι η παράδοση των γυναικών είναι η αντίσταση και θεωρώ ότι

Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τη Λέλα Γκιουβέν για τον αγώνα της, για τη θυσία της. Την υποστηρίζουμε, την κατανοούμε. Οι συνάδελφοι τώρα θέλουν το λόγο, παρακαλώ. Πολύ σύντομα όμως, παρακαλώ. Γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Γυναικών που αποδέχθηκε το αίτημά μας να έρθει εδώ η Τέιλα Γκιούβεν. Πρόκειται πραγματικά για μια σημαντική μαρτυρία την οποία ακούσαμε σήμερα. Ακόμα και αν η Λέιλα δεν μπορούσε να είναι εδώ μαζί μας. Να προσθέσω και να θυμίσω κάποια πράγματα. Η Λέλα Γκιουβέν απεργεί, κάνει απεργία πίνης από τις 8 Νοεμβρίου του 2018 για να και ζητάει να σταματήσει η απομόνωσή τη. Υπάρχουν πολλοί όμως άλλοι Κούρδοι οι οποίοι είναι σε απεργία πίνας και όλοι μας ζητούν να ακουστεί η φωνή αυτή να μιλήσουμε επιτέλους στην Ευρώπη και να δράσουμε στην Ευρώπη όχι μόνο κατά της απομόνωσης του Οτσαλάν, αλλά και κατά της συνεχούς παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Κάτι το οποίο φάνηκε και τώρα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι η Επιτροπή Γυναικών ε, να παίζει αυτό το ρόλο. Θα το πω και θα το λέω πάντα. όχι μόνο επειδή το κουρδικό ζήτημα είναι πολύ σημαντικό για μας ε, και για μένα, εγώ αισθάνομαι και υπόχρεη απέναντι στις γυναίκες του Κουρδιστάν για αυτό που εκπροσωπούν. Μας έδειξαν πώς μπορούμε να σκεφτούμε αλλιώς την πολιτική από την πλευρά των γυναικών, από τη δύναμη των γυναικών που δίνουν έναν αγώνα κατά του ISIS. Νομίζω ότι πραγματικά χρωστάμε σε αυτές τις γυναίκες θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε αυτό το χρέος να το αποπληρώσουμε τουλάχιστον υποστηρίζοντα τη Λεϊλά Γκιουβέν. Ελπίζω λοιπόν η Επιτροπή μας και όλες από εμά σε αυτούς τους δύο μήνες της εκστρατείας, όλες μας, στα κράτη-μέλη μας, θα κάνουμε κάτι και σε ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και άλλη μια φορά τις γυναίκες από το Κουρδιστάν. Παρακαλώ, η κυρία Μπιόρκ έχει το λόγο. Να ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω θερμά τις φίλες που ήρθαν εδώ. Θέλουμε να στείλουμε το τους χαιρετισμούς μας στη Λέιλα Γκιουβέν. Βεβαίως η Λέιλα Γκιουβέν εκπροσωπεί είναι μια πολύ σημαντική πολιτική προσωπικότητα. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνει βέβαια η απεργία πείνας. Εδώ μιλάμε για την Επιτροπή Γυναικών και είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να ακουστεί αυτή η φωνή εδώ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, για την ελευθερία, για την καταπολέμηση ενό αυταρχικού αντιδημοκρατικού καθεστώτος όπως αυτό του κ. Ερντογάν. Εγώ συνάντησα στο Στρασβούργο μια γυναίκα που κάνει απεργία πείνα και μου είπε το εξή: Όταν κάποιο βρίσκεται απέναντι στο φασισμό, πρέπει να κάνει κάτι. Όταν πια δεν μπορεί κανεί να διαδηλώσει δεν μπορεί καν να εκφράσει την άποψή του, να συζητήσει. Δεν μπορεί να εργοτράσει ως δημοσιογράφος. Δεν μένουν και πολλά πράγματα, δεν μένουν και πολλά όπλα. Πέρα λοιπόν από την υποστήριξη στον αγώνα σας, θα πρέπει να μας πείτε κι εσείς τι θέλετε από μας, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για σας, διότι όλοι όσοι δίνουν αυτή τη μάχη, όλοι όσοι ε, μάχονται για τη δημοκρατία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, πρέπει να ξέρουν ότι είμαστε στο πλάι τους. Δεν είναι μόνο η Λέιλα, είναι εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι που βρίσκονται στη φυλακή για πολιτικούς λόγους. Είναι δηλαδή πολιτικοί κρατούμενοι που διακυβεύουν τη ζωή τους. Στον αγώνα που δίνουμε για μια ευρωπαϊκή Τουρκία αλλά και μια δημοκρατική Τουρκία αλλά και μια δημοκρατική Ευρώπη ε, θέλουμε να μας πείτε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε. Είμαστε ευρωβουλευτές, ε, μπορούμε να κάνουμε κάτι κι εμείς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και στείλτε τα χαιρετίσματά μας τα πιο θερμά στη Λέιλα. Θα είμαι σύντομη διότι έχω ήδη μια πολύ καλή συνεργασία με τις γυναίκες του Κουρδιστάν. Ήμουν στον Τιγερμπακύρ τον Ιανουάριο με τη Ματίνα Άντερσον. Προσπαθήσαμε εκεί παρέμβουμε ζητώντας την άδεια να δούμε τη Λέλα Γκιουβέν που ήταν στη φυλακή δεν μας έδωσαν την άδεια αυτή όμως μετά από λίγες μέρες την απελευθέρωσαν νομίζω λοιπόν ότι τέτοιες παρεμβάσεις πιάνουν τόπο και κάτι μπορούν να αλλάξουν όταν δρούμε από κοινού είναι πραγματικά πολύ σημαντικό ότι βρίσκεστε εδώ σήμερα και ότι βρίσκεστε στο πάνελ αυτό, διότι συχνά τα θέματα για τα οποία συζητάτε ε, θεωρούνται πολύ περίπλοκα ε, και τα αφήνουμε στο περιθώριο. Ε, πραγματικά είμαι περήφανη που είστε εδώ σήμερα. Είμαι περήφανη που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μέρος όπου το Λαϊκό Δικαστήριο έδωσε την τιμιγορία του, ε, την του στον αγώνα του κουρδικού λαού απέναντι στην Τουρκία. Έγινε εδώ αυτή η διάσκεψη, αυτό το, αυτή η δίκη στο Ευρωπαϊκό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δίνουμε τη μάχη μαζί σας. Βεβαίως και πρέπει να επικρίνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει και να την ε, συγχαρούμε αυτή τη σημαντική πλατφόρμα που αποτελεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ορισμένε φορέ υπάρχει μια σύγχυση όταν μιλάμε για την Ευρώπη. Πρέπει να επικρίνουμε ίσω περισσότερο το Συμβούλιο. Διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιοι βεβαίω είναι στην λαθασμένη πλευρά, αλλά εσεί είστε εδώ σήμερα. Ερχόμαστε και στι φυλακέ ε, να σα δούμε. Οργανώνουμε συνεντεύξει τύπου, διασκέψει Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί αυτή η φωνή. Α εξασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε από αυτού. Ξέρετε, και εγώ έδωσα μάχη για τη Λέιλα Μπάρεκ όταν ήταν φυλακή. Ε, ίσως ε, να είναι κάτι πρακτικό που μπορούν να κάνουν γυναίκες ευρωβουλευτίνες ε, σε αυτές τις περιπτώσεις στέλνοντας επιστολές, κάρτες, πολλές και διάφορες δράσεις όπου λέμε ότι ξέρετε υπάρχει κάποιο ο οποίος έχει εκλεγεί βουλευτή, όπω και εγώ και αυτό είναι στη φυλακή και εγώ δεν είμαι και εγώ την υποστηρίζω. Είναι εξαιρετικά συγκεκριμένο και πρακτικό αυτό νομίζω. Ευχαριστώ πολύ. Ε, την απάντησή σας λοιπόν.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 Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, συμβολή σας και για τα σχόλιά σας και θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά που μας δώσατε τη δυνατότητα να εκφράσουμε την, ε, ε, την Λέιλα Γκιουβέν και να αποτελέσουμε τη φωνή της εδώ όπως και η Margaret Owen ας πούμε ε, που είναι πολύ ε, γνωστή ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε απεργία πείνας σήμερα στο Λονδίνο για να δείξει την αλληλεγγύη της προς την Λεϊλά. Είναι 75 χρονών, δικηγόρος και συγγραφέας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 ότι πάντα υπάρχει διασύνδεση ανάμεσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά ε, όργανα και ε, τους θεσμούς στην ε, Τουρκία. Έχετε επαφές μαζί τους και επομένως θα μπορούσατε ίσως να ασκήσετε πίεση μέσω των κυβερνητικών οργανώσεων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που μια αντιπροσωπεία προσπάθησε να επισκεφθεί την Λέιλα και ε, ε, ε, η πνευματική εγκύτητα επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως μπορείτε να στείλετε και κάποια αντιπροσωπεία για να δείτε ποια είναι η κατάσταση των φυλακισμένων στην Τουρκία. και ό,τι μπορείτε να κάνετε για να σταματήσουν οι θάνατοι στις φυλακές. Ξέρετε ότι Εφτά ε, νέοι Κούρδοι ε, αυτοκτόνησαν στις τουρκικές φυλακές ε, έτσι ώστε να επιστήσουν την προσοχή του κόσμου στο θέμα αυτό. Είναι πολλές οι κινήσεις κατά της δημοκρατίας στην Τουρκία και είμαι σίγουρη ότι κάτι θα βρείτε να κάνετε έτσι ώστε να σταματήσετε την κατάσταση αυτή. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό λοιπόν να σας πω ότι ε, ε, μπορείτε να ασκήσετε πίεση για το ε, CPT. Αυτά ήθελα να πω για την ώρα. Σας ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά που μας δώσατε αυτή τη δυνατότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Οπωσδήποτε υποστηρίζουμε την Ελέηλα αλλά και την κουρδική κοινότητα στο σύνολό της ε, που αγωνίζεται για την ελευθερία. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε με το σημείο υπαριθμών 6 που είναι η αποστολή στην ε, Ισπανία. Ε, δεν έχουν υποβληθεί σχόλια σχετικά με την έκθεση για την αποστολή αυτή και επομένως ε, την εγκρίνουμε την έκθεση και φτάνουμε στο σημείο υπαριθμών 7 που αφορά τον διάλογο με τις ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις όσον αφορά διάφορες, διαφορετικές μορφές διακριτικής μεταχείρισης θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά αυτό το θέμα αυτό και ε, χρειαζόμαστε λίγο χρόνο έτσι ώστε οι εμπειρογνώμονες εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων να πάρουν τη θέση τους στο πάνελ. E, e, Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα ε, στον ε, ε, υπεύθυνο για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Φασισμού, στην υπεύθυνο μάλιστα, την κυρία Ιζαμπέλα Ευχαριστώ πάρα πολύ. Του ρατσισμού, συγγνώμη. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τον λόγο. Σαν γυναίκες μερικές φορές ε, πρέπει να κάνουμε μόνες μας πράγματα. Ας πούμε έχουμε... Ε, ε η, η συνάδελφος έπρεπε να πάρει το παιδί της από τον παιδικό σταθμό, γι' αυτό μοιράσαμε λίγο την παρουσίαση. Ζητώ την κατανόησή σας. Θα προσπαθήσω ε, να αναφερθώ και στα δύο ε, τμήματα. Ε, εγώ, ενώ τα είχαμε χωρίσει, θα πρέπει να μιλήσω και για τα δύο. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να μην φανεί σαν σειραφή. Θα ξεκινήσω με αυτά που εγώ θα έλεγα ε, καταρχήν. Τι εννοούμε δηλαδή με αυτήν την έννοια της intersectionality, αυτής της πολλαπλότητας. Ε, μιλάμε για ε, διάκριση που αφορά και το φύλλο και την σεξουαλική, το σεξουαλικό προσανατολισμό και τον ε, την θρησκεία κλπ. Δηλαδή ε, πολλαπλές μορφές διάκρισης και πώς αυτές ε, μπορεί να επηρεάσουν το άτομο. Σε πολλές καταστάσεις ε, μπορεί μια γυναίκα να υποστεί διακριτική μεταχείριση όσον αφορά τον, ε, την αναπηρία της, ε, το κοινωνικό της καθεστώς, το καθεστώς της ως πρόσφυγα ή μετανάστριας κλπ. Όλες αυτές οι αρχές δημιουργούν ένα μεγάλο χάσμα και μπορεί να οδηγήσουν ε, σε μεγάλες διακρίσεις ε, ε, ας πούμε για μαύρες πρόσφυγες ή για γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν και τη φτώχεια και είναι μέλη της LGTB κοινότητας κλπ. Ε, η κοινωνική συμπερίληψη λοιπόν είναι αυτή η οποία θα πρέπει να ε, ε, επιδιώκεται πέρα από οποιοδήποτε άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ας πούμε αν είναι μια γυναίκα μαύρη ή αν ανήκει στους Ρωμά όπως και εγώ η ίδια. Ε, γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν τέτοιες πολλαπλές ε, συνθήκες ε, μπορεί να αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης πολύ πιο συχνά. Και θα ήθελα να περάσω τώρα στο επόμενο σημείο που είναι η αντιμετώπιση της από πλευράς του νόμου. Αλλά πριν από αυτό να αναφερθώ σε μία υπόθεση η οποία ονομάζεται The Grand Ferrite όπου στην General Motors στο ε, Μιζούρι οι γυναίκες είχαν ε, διαφορετική αντιμετώπιση. Σύμφωνα όμως με την αρχή ε, της ε, ισότητας ε, το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πρόβλημα γιατί για τις λευκές υγιείς γυναίκες δεν υπήρξε διαφορετική αντιμετώπιση από τους λευκούς υγιείς άντρες. Ωστόσο υπήρξε διακριτική μεταχείριση όσον αφορά άλλες γυναίκες. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει συγκεκριμένο πεδίο που να αντιμετωπίζει, πλαίσιο συγγνώμη, για την αντιμετώπιση των πολλαπλών ε, ταυτόχρονων ε, διακρίσεων. Υπάρχουν ε, όμως μονάχα κάποιες αιτιολογικές σκέψεις χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα. Ε, μονάχα ε, μπορούμε να αναφέρουμε νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτρέπουν ή απαγορεύουν την διάκριση ε, λόγω φύλου ή λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή προστασία όσον αφορά τις γυναίκες για το μισθολογικό χάσμα, για τις άδειες για, το, για την εγκυμοσύνη, την περίοδο γαλουχίας, τη κοινωνική ασφάλιση κλπ οι πολλαπλές διακρίσεις ή intersectional discrimination δεν αναφέρονται ε, συγκεκριμένα στο ευρωπαϊκό, στο, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Απλώς αναφέρεται ε, μια γενική αναφορά ε, σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες θα πρέπει ιδιαιτέρως να προστατεύονται μια και πολύ συχνά αποτελούν αντικείμενο πολλαπλών διακρίσεων. Αλλά αυτό αναφέρεται στις διάφορες μορφές διάκρισης και όχι στην ταυτόχρονη ύπαρξη πολλαπλών ε, διακρίσεων. Κατά την άποψή μου λοιπόν, τα κράτη-μέλη θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουν αυτήν την intersectionality, την ταυτόχρονη πολλαπλή, δηλαδή ε, ε, την ύπαρξη ταυτόχρονα πολλών παραγόντων διάκρισης. Ας πούμε, εάν μία βορειοαφρικανή ε, γυναίκα θέλει να ενοικιάσει σπίτι, πρέπει να της το νοικιάσει κανείς, αλλά ε, δεν ε, δημιουργείται πρόβλημα εάν αυτή η γυναίκα δεν τελικά νοικιάζει το διαμέρισμα, δεν της το νοικιάζουν λόγω της θρησκείας. Γιατί η θρησκευτική ελευθερία διασφαλίζεται μονάχα στο χώρο της δουλειάς. Επίσης ε, δεν προβλέπονται θετικές ε, ε, δραστηριότητες ή δράσεις κατά την ίδια έννοια. Επίσης, στο Συμβούλιο δεν έχουν προχωρήσει τέτοιου είδους διατάξεις γιατί απαιτούν ομοφωνία. Δεν υπάρχει λοιπόν πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόθεση του, αντι, του νόμου κατά των διακρίσεων, ωστόσο η, παρόλα αυτά, ε, η υπομαλτέζικη προεδρία ε, προώθησε, προχώρησε λίγο το θέμα της διακριτικής μεταχείρισης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό η Ευρωπαϊκή Κοινωνική ε, και Οικονομική Επιτροπή επίσης έχει ε, κάνει γνωμοδοτήσεις ε, σχετικά με το θέμα αυτό και σχετικά συγκεκριμένα με την intersectionality. Εμείς ε, ε, θεωρούμε ότι ε, υπάρχει νομοθεσία κατά της διακριτικής μεταχείρισης, αλλά που κάθε φορά αφορά μία συγκεκριμένη μορφή διάκρισης, ενώ εμείς πιστεύουμε ότι η ύπαρξη πολλών ταυτόχρονων στοιχείων δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα και ε, επίσης ε, θεωρούμε ότι ε, λόγω της ύπαρξης πολλαπλών μορφών διάκρισης ή στοιχείων μάλλον διάκρισης δημιουργείται μια διαφορετική δυναμική η οποία μπορεί να δημιουργήσει στο σύνολο μεγαλύτερη απομόνωση. Επομένως θα πρέπει να δούμε γυναίκες ας πούμε ε, λευκές ε, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω του χρώματος αλλά λόγω του φύλου τους οι μαύρες γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω του χρώματος του δέρματός τους αλλά και λόγω του γεγονότος ότι είναι γυναίκες. Single identity Επομένως, ε, το ε, ε, κεντρικό πρόβλημα αυτής της intersectional discrimination είναι πώς μπορεί κανείς να νομοθετήσει έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα πολλαπλά μειονεκτήματα. Νομίζω ότι θα πρέπει καλύτερα να καταλάβουμε την ίδια την έννοια, την ουσία της διάκρισης, γιατί αυτά αυτές οι ομάδες δεν είναι ποτέ ε, ομοιογενείς και η ιεράρχηση των ομάδων ή η ιεραρχία εντός των ομάδων ποτέ δεν είναι ε, ίδια. Ε, προκαλείται όμως πάντοτε πολλαπλός αποκλισμός λόγω ακριβώς των συγκεκριμένων μορφών διάκρισης που βασίζονται είτε στην εθνοτική, είτε σε εθνοτικά στοιχεία, είτε σε θρησκευτικά, είτε σε σεξιστικά κλπ χρειάζονται οπωσδήποτε πιο αποτελεσματικά μέτρα ε, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στο σύνολό τους. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ε, την αλληλεγγύη έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε την ισότητα. Η διακριτική μεταχείριση μπορεί να βρίσκεται σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορα πεδία και επομένως χρειάζεται συνολική αντιμετώπιση. Πρέπει να ξεπεράσουμε την αντίληψη της ισότητας που βασίζεται μονάχα ε, στην αρχή ότι ε, θα πρέπει παρόμοια στοιχεία να αντιμετωπιστούν με παρόμοιο τρόπο. Ε, η ισότητα θα πρέπει να συμπεριλάβει περισσότερες διαστάσεις. Ε, θα πρέπει να ξεπεραστούν τα στερεότυπα, η βία, ε, ο στιγματισμός. Θα πρέπει να διευκολυνθεί, να ακουστεί η φωνή των ανθρώπων που έχουν υποστεί διακριτική μεταχείριση. Επίσης, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις πηγές διακριτικής μεταχείρισης σε διαφορετικά περιβάλλοντα καθώς επίσης χρειαζόμαστε και ε, κεντρικά μέτρα τα οποία θα αντιμετωπίσουν όσο γίνεται ε, περισσότερες ομάδες. Σε επίπεδο ε, κρατών χρειαζόμαστε κράτη τα οποία θα λαμβάνουν κεντρικά μέτρα έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η πολλαπλή διάκριση. αυτή η intersectionality θα πρέπει να ξεπερνάει ε, ή μάλλον να είναι μια εγκάρσια πολιτική ε, στα προγράμματα ε, κατά των διακρίσεων που μπορεί να έχουν τα διάφορα κράτη και εκτός από την πολιτική ισότητα να αναλαμβάνουν και δράση όσον αφορά αυτήν την intersectionality, την πολλαπλή διακριτικότητα ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε και ποια είναι τα στοιχεία. Ε, ε, υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετά στοιχεία τα οποία μπορεί να συλλεγούν και να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε ε, να δημιουργηθούν ε, περισσότερο, να, να, να οικοδομηθεί γνώση όσον αφορά αυτές τις ομάδες. Θα πρέπει να υπάρχει ε, και ε, μια έκθεση ανά πενταετία έτσι ώστε ε, να έχουμε λεπτομερείς πληροφορίες καθώς επίσης και επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με οποιαδήποτε διάκριση από οποιαδήποτε πηγή και σε οποιαδήποτε μορφή. Στρατηγικό σχεδιασμό έτσι ώστε να βελτιωθεί η στρατηγική που θα βασίζεται πλέον στην intersectional analysis. Νομίζω επίσης ότι και εσείς σαν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να απαιτήσετε ε, να ε, ε, συμμετοχή στο θέμα αυτό και επομένως να εκπονήσετε ψήφισμα κατά την έννοια αυτή έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι δεν θα ξεχαστεί αυτή η συζήτηση για την intersectionality. Άρα, είσαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή ε, να αντιμετωπίσετε αυτή την πρόκληση. Ελπίζω να μην ήμουν ακατανόητη, γιατί προσπάθησα να σειράψω δύο διαφορετικές... Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν πολύ επιτυχή σε αυτή την προσπάθεια. Ποιος θα θέλει να πάρει το λόγο, μάλλον. Μάλιν Μπιόρκ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω στο ειδικά. Αυτοί που ανήκουν στην ε, αριστερά κάνουν λόγο πάντα για αυτό το θέμα της διατομιακής διακριτικής μεταχείρισης. Για πολλούς ανθρώπους, ε, διάφορες περιστάσεις που υποφέρουν από αυτή τη διακριτική μεταχείριση. Μας δείξατε τη δικιά σας οπτική και θεωρώ ότι θεωρώ ότι αυτή είναι η Επιτροπή που διαρκώς κάνει αναφορά σε αυτό το θέμα. Βέβαια, ε, σε άλλες επιτροπές δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε και πολλά πράγματα. Υπάρχουν διαφορετικοί τομείς και συγκεκριμένοι τομείς όπου κάναμε λόγο για τη διάκριση των ε, γυναικών. Κάναμε λόγο για τις διαφορετικές μορφές διακριτικής μεταχείρισης ενάντια των γυναικών, εις βάρος των γυναικών, εξαιτίας της εθνικότητάς τους, του γεγονότος ότι βρίσκονται σε φυγή. Και πάντα λέγαμε ότι αυτή η διατομική διακριτική μεταχείριση ως έννοια λείπει έχει να κάνει με διακρίσεις εξαιτία διαφορετικών λόγων όπως είναι ο ρατσισμός και υπάρχουν και τομείς που έχουν να κάνουν με το ρόλο της γυναίκας, την ριζοσπαστικοποίηση νέων και αυτό μου θυμίζει την ριζοσπαστικοποίηση των γυναικών ε, στο Ισλάμ όπου θα μπορούσαν να, να λειτουργήσουμε προληπτικά και φυσικά αυτό θα μπορούσαμε να το μεταφέρουμε και σε, άλλους, ε, σε άλλες μορφές τρομοκρατίας. Υπάρχει βέβαια και παράλληλα πολύ μεγάλη απειλή από ακροδεξιές δυνάμεις και αυτό είναι ένας κίνδυνος που δεν έχουμε λάβει ε, αρκετά σοβαρά σε αυτή την Επιτροπή. Και φυσικά θα πρέπει να αποτελέσει μια πρόκληση για εμάς, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες γυναικών που αντιμετωπίζουν αυτού του είδους τη διάκριση, που στιγματίζονται επίσης και θεωρώ ότι η εποχή μας είναι άκρος ρατσιστική. Θα πρέπει να αγωνιστούμε για τα δικαιώματα όλων των γυναικών, αλλά σε διάφορους τομείς. Όπως είπατε, είναι νομικό το θέμα. Όμως δεν αρκεί μονάχα να υιοθετήσουμε νομοθεσίες. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να περισπαστούμε τα δικαιώματα των γυναικών. Έχουμε προετοιμάσει μία πρόταση τροπολογίας για μια απόφαση του δικαστηρίου όπου δίνεται το δικαίωμα στον εργοδότη να ε, διακρίνει τις γυναίκες με το αν φοράνε κάποιο μαντήλι, κάποια μπουρκα ή οτιδήποτε σχετικό. Είναι μια απόφαση που ε, στοχεύει ακριβώς τις μουσουλμάνες. Από την πλευρά των αριστερών κάναμε μία πρόταση τροπολογία και ασκούμε κριτική σε, αυτό, σε αυτή την απόφαση τη δικαστική. Δεν καταφέραμε και πολλά. Δεν έχει επομένω να κάνει μόνο με τις δικαστικές αποφάσεις, αλλά και με τις δικέ μας προσπάθειες ε, στο να συμπεριλαμβάνουμε στι εκθέσεις μας ε, αυτή την πτυχή για τη δικαίωμα των γυναικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες να καταπολεμήσουν τον ρατσισμό, πώς μπορούμε να κάνουμε ως ε, παράγοντες, ως ε, κοινοβούλιο. Αυτό το θέμα της ε, διαδομιακής διακριτικής μεταχείρισης έχει να κάνει με ανθρώπους ναι με, αλλά από πλευρά πολιτικής το ερευνούμε γιατί είναι δύσκολο να έχουμε συγκεκριμένες ε, διακρίσεις σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων όπως είναι οι μουσουλμάνες γυναίκες, οι γυναίκες Ρώμα, ε, οι μαύρες γυναίκες. Δεν έχει αναγνωρίσει συγκεκριμένες ε, διακρίσεις όπως θα έπρεπε, όπως η φοβία για τους μουσουλμάνους κτλ. δεν έχουμε τη δυνατότητα και από νομικής πλευράς να ε, καταπολεμήσουμε την, την διατομική διακριτική μεταχείριση. Υπάρχουν δύο τρόποι να το πράξουμε. Σε επίπεδο πολιτική και νομοθεσία. θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις συγκεκριμένε μορφές ρατσισμού, να τις ονοματίσουμε, να τις ορίσουμε Έχουμε ένα ψήφισμα για γυναίκε αφρικανική καταγωγή, αλλά θα πρέπει να το κάνουμε αυτό και για άλλε κατηγορίε γυναικών, για τι μουσουλμάνε π.χ. Και παράλληλα θα πρέπει να δούμε την διατομεακή πτυχή ω νομική έννοια και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, γιατί σε εθνικό επίπεδο είναι δύσκολο να έχουμε ε, Διατάξει που να αφορούν την διατομιακή διακριτική μεταχείριση. Όσον αφορά τη συμπερίληψη των γυναικών αυτών, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ομάδε εργασίε εντό του Κοινοβουλίου όπου θα κάνουμε λόγο για τον, τον αντίκτυπο ποιοι τη Ισλαμοφοβία στι μουσουλμάνε γυναίκε. Έχουμε ένα σχετικό φόρουμ αύριο και να δημιουργήσετε το χώρο για να μπορούν να έρχονται εδώ και να σα απευθύνουν το λόγο για να γνωρίζετε πώς μπορείτε να προχωρήσετε σε, το, ε, σε τροπολογίες, πώς θα αποτρέψετε την ριζοσπαστικοποίηση. Γιατί δυστυχώς αυτό που σημαίνει πολλές φορές είναι ότι όταν δεν εμπλέκουμε στη διαδικασία στις γυναίκες οι οποίες πλήττονται από τέτοια θέματα εξτρεμισμού, τότε υιοθετούμε τη λάθος νομοθεσία, προτείνουμε λάθος τροπολογίες. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τις προστατέψουμε τις γυναίκες αυτές που είναι θύματα βίας και ζωσπαστικοποίησης. Ναι, με το ψηφίσμα εγκρίθηκε, αλλά θα πρέπει να εμπλέξουμε την κοινωνία των πολιτών, να οργανώσουμε ακροάσεις, ομάδες εργασίας, για να συνεχιστεί και αυτή η δουλειά και στην επόμενη θητεία. Να δούμε τι μπορεί να γίνει μέσα στο τρέχον πλαίσιο. Να υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που θα ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα, όπως μουσουλμάνες, γυναίκες Ρώμα, γυναίκες αφρικανικής καταγωγής κτλ. Ε, μετανάστριες κτλ. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε και επίσης να γίνεται και σε εθνικό επίπεδο προσπάθεια για την ε, ενδυνάμωση των γυναικών, την κατάρτιση των γυναικών, για την εμπλοκή τους στις πολιτικές. Όλο και περισσότερο. Πόσοι Ρώμα έχουμε στο Κοινοβούλιο, πόσες Αφρικανικής καταγωγή θα έχουμε στην επόμενη Βουλή, πόσε Μουσουλμάνες εδώ στην επόμενη μου Όλα αυτά πρέπει να τα αναλογιστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Συμφωνούμε βεβαίω. Πρέπει να συνεργαστούμε και θα πρέπει να συμμετέχουν και η ΜΚΟ, η κοινωνία των πολιτών για να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις για να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι ε, πολλαπλέ μορφέ ε, διακρίσεων. Σα ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα εδώ. Συνάδελφοι, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Περνάμε στο σημείο 8 τη ημερησία διάταξη, Το σχέδιο δράση ε, για τα δύο φύλλα. Η αντιπροέδρο του Κοινοβουλίου, η κυρία Γκέπχαρτ, είναι εδώ για να μα μιλήσει γι' αυτό. Παρακαλώ. Κυρία Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Εκπροσωπώ τον πρόεδρό μας του, της ομάδας υψηλού επίπεδου. Είμαι μέλος της ομάδας αυτής και φυσικά ασχοληθήκαμε εντατικά με την έκθεση της κυρίας Νινά. Στη σημερινή συνεδρίαση θα συζητήσουμε αυτά που θέλουμε να εφαρμόσουμε και που περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση. Είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση και θέλω να καταστήσω σαφές εδώ ότι στο Προεδρείο σε κάθε συνεδρίαση έχουμε το θέμα της ισότητας στην ημερήσια διάταξη. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το θίγουμε συνεχώς, διαρκώς και πάντα θέλουμε να ενημερωνόμαστε για τα πεπραγμένα Θέλουμε να εξετάζονται όλες οι προκηρύξεις για θέσεις εδώ στο Κοινοβούλιο και αν τηρούνται οι κατάλληλες αναλογίες στο θέμα το... της ισότητας των φύλων. Στη Στουτγκάρδη, στο Έσμπαν, είδα μία αγγελία για θέσεις και εκεί είχε τρία φύλλα. Κάνα αναφορά σε τρία φύλλα, όχι σε δύο. Και πάντα υπάρχουν τέτοια θέματα τα οποία πρέπει να σκεφτόμαστε. Και όταν αλλάζουν οι προκηρύξεις, πάντα βλέπουμε αν έχουν γίνει σωστά. Θα ήθελα να σας πω όλα αυτά που έχουμε κάνει, όμως έχουμε λίγο χρόνο και γι' αυτό το λόγο θα, θα εστιάσω σε τρία σημεία που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα αφήσω στην άκρη το πακέτο που έχω. Δύο σημεία ειδικά όσο όπως είναι η της πρωτοβουλίας της κυρίας Νίνα στο σημείο 17 θα μιλήσουμε αύριο για ένα έγγραφο στο συστημα ψηλού επίπεδου Θα έχουμε τη αύριο στο Προεδρείο το απόγευμα για να αποσαφηνίσουμε αυτές τις, ε, αυτά τα αιτήματα και έχουμε πρόθεση το σημείο 17 να το ε, καθιερώσουμε Επίσης θα πρέπει να υπάρχει εποπτεία στην εφαρμογή. Θα πρέπει να διοριστεί όμω κάποιος για να αναλάβει αυτό το πόστο. Αυτό δεν το περιλαμβάνουμε στην έκθεση, αλλά γνωρίζουμε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι καλές, αλλά εφαρμόζονται σωστά μόνο όταν υπάρχει εποπτεία. Αν συμφωνήσετε, θα προτείνω ε, κάτι που δεν περιλαμβάνεται στην έκθεση, αλλά που κατά την άποψή μου είναι σημαντικό. Γίνεται λόγος ε, για την διοίκηση του Ευρωκοινοβουλίου που θα πρέπει να είναι προσεκτικές προς το θέμα αυτό. Αυτό θα το απευθύνω και για τα κόμματα, γιατί και στα κόμματα, στις πολιτικές ομάδες υπάρχει διοίκηση και θα πρέπει και αυτά να λάβουν υπόψη αυτό το, το θέμα. Στα σημεία 24α ω C, η αρμόδια επιτροπή πρότεινε όλα τα μέλη του Ευρωκοινωνίου να περάσουν από μια εκπαίδευση αλλά μόνο αυτά τα μέλη που θέλουν να εκπληρώσουν ε, κάποια, ε, κάποιο ρόλο στο κοινοβούλιο. Νομίζετε ε, και τι εκπαιδεύσει που γίνανε ενάντια στην παρενόχληση κτλ. Γίνανε σε αυτή τη θητεία και στο επόμενη, στην επόμενη θητεία θα γίνουν. Ε, τις ψηφοφορίες δυστυχώς τις χάσαμε σε σχέση με αυτό το θέμα. Όμω παραμένει ένα θέμα το οποίο θέλουμε να προωθήσουμε και στο μέλλον και είναι πολύ σημαντικό να φροντίσουμε να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι θα πρέπει να κάνουν λόγο για τις ανεπιθύμητες πράξεις, τις σεξουαλικές παρανοχλήσεις και θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Η Αρμόδια Επιτροπή για την Παρενόχληση έρευνα τη δημιουργία μιας ομάδας με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Η πλειοψηφία θεώρησε ότι θα ήταν καλύτερα να γίνουν όλα εσωτερικά. Όμως θεωρώ ότι η άποψη των εμπειρογνωμών, κοινωνιολόγων και ψυχολόγων θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Το ζήτησε και η Ευρωπαία Διαμεσολαβητή σε μία πρόταση τη 17 η Δεκεμβρίου του 2018. Έχουμε κάνει κάποιε πρόταση στο Κοινοβούλιο. Θα ήταν όμω ε, λάθος να ε, αρκεστούμε σε αυτό. Γιατί δεν θα είχαμε πετύχει τίποτα αν δεν ε, αν Και στο Προεδρείο, άλλη μια φορά θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό την επόμενη εβδομάδα. Βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε, αλλά η Μογάν Σαρτιέ, η, η απεργούσε. Οπότε θα το ε, δούμε στην επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Γκέπχαρτ που ήρθε στην Επιτροπή μας. Να σας ευχαριστήσω και για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης αυτού. Έχετε ρωτήσει, συνάδελφοι, σχόλια για την κυρία Γκέπχαρτ. Παρακαλώ, η κυρία Νόιχελ. Äh, στην Επιτροπή ΦΕΜ Κάνουμε λόγο για δύο πράγματα. Τα γνωρίζεις ήδη, αλλά είναι σημαντικό να τα τονίσουμε. Σημαντικό είναι ότι όλοι που έχουν ευθύνη για το προσωπικό, άντρες και γυναίκες, να περάσουν εκπαίδευση για το θέμα της σεξουαλικής περνόχλησης, του εκφοβισμού είναι μια, ένας συμβασμός να πούμε ότι ναι, δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τους πάντε να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση αυτή. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είναι υποχρέωση για όλους. Το δεύτερο έχει να κάνει με τους εξωτερικού εμπειρογνώμονε. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα συστήματα, είτε είναι η Καθολική Εκκλησία, είτε το Ευρωπαϊκό έχουν Ε, φροντίζουν για ορφανοτροφία, τα οποία έχουν εσωτερικές, εσωτερικά προβλήματα και στα οποία μπορούν να βρεθούν πολύ καλές λύσεις από έξω. Ακόμα και η Καθολική Εκκλησία προσπάθησε εσωτερικά να βρει τρόπους και το Ευρωκοινοβούλιο, όμως δεν ήταν επαρκές. Ήταν λίγα αυτά που έγιναν. εκεί όμως που υπάρχουν ε, θέματα υπάρχουν επιθέσεις πάντα σε καθημερινή βάση και θα ήταν κρίμα ότι κάποιοι πιστεύει ότι θα είναι στίγμα για το Κοινοβούλιο να ασχοληθούμε πιο εντατικά με αυτό το θέμα. Δεν είναι λάθος να πούμε ότι υπάρχουν λάθος συμπεριφορές. Το να πούμε σε συναδέλφους ότι τη συμπεριφορά σου δεν ε, την αποδέχουμε. Το λάθος είναι να αποσιωπούμε και να συγκαλύπτουμε τέτοιες καταστάσεις. Ένας Πολωνός βουλευτής κατάφερε να γλιτώσει όταν είπε ότι είναι δίκαιο οι γυναίκες να παίρνουν χαμηλότερους μισθούς. Το θεωρώ απαράδεκτο, σεξιστική δήλωση. Και τελικά δεν του επιβλήθηκε κάποια ποινή για αυτή τη δήλωση. Σε ευχαριστώ, Εύελιν, που αγωνίζεις για αυτό το θέμα. Όμως πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα. Δεν έχουμε πετύχει αρκετά. Ευχαριστώ ο κ. Ευχαριστώ την κυρία Γκέπχαρτ που είναι εδώ μαζί μας. Δύο-τρία θέματα θέλω να θίξω. Πρώτα απ' όλα θα προτείνετε το Προεδρείο να εγκρίνει κάτι πριν το τέλος της θητείας. Θα υπάρξει απόφαση για το σχέδιο δράση το Προεδρείο. Θα υπάρχει τέτοια σύσταση από την πλευρά σα. Διότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Και κάτι άλλο που δεν ξέρω τι θα κάνετε εσεί. Να γίνει μια εξωτερική αξιολόγηση για το τι συμβαίνει στο Κοινοβούλιο. Διότι έχουμε διάφορα όργανα. Ε, η Επιτροπή ΦΑΜ με, το ετήσιο, με την ετήσια έκθεση, ε, οι υπηρεσίε έρευνα που κάνουν σχετικέ μελέτε, μια εξωτερική όμω ε, έρευνα που θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Γυναικών για όλα αυτά τα θέματα ε, θα ήταν χρήσιμο. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί κάτι τέτοιο. Επίσης, σε σχέση με αυτό που είπατε για την ε, σεξουαλική παρενόχληση των μελών, είπατε ότι χάσαμε την ψηφοφορία ε, την προηγούμενη φορά. Άλλε φορέ την έχουμε κερδίσει όμω. Δεν ξέρω πότε μπορεί να το επαναφέρετε το θέμα πάντω και για την ομάδα υψηλού επίπεδου. Ε, Μήπω υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Πάντω το βασικό που θέλω να πω είναι ότι εφόσον είμαστε στο τέλο τη θητεία, να αφήσουμε κάτι συμφωνημένο στο Προεδρείο. Έτσι. Είναι το ελάχιστο νομίζω που πρέπει να προσπαθήσετε να κάνετε. Äh, Ευχαριστώ. Θα σας δώσουμε κάτι εγγράφος. Δεν θέλουμε η δουλειά πέντε χρόνια πάει στράφη. Θα υπάρξουν έγγραφα και αποφάσεις και όσον αφορά την εκπαίδευση και τα βήματα στα οποία έκαναν αφορά θα είναι και αυτά αποφάσεις, όχι συστάσεις για τη διοίκηση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ήταν πολύ προβληματικό το αντίθετο. Αύριο στην ομάδα ψηλού επίπεδου θα το αποφασίσουμε αυτό και θα έχουμε ένα άρθρο 228 για το ζήτημα αυτό. Επίσης, όσον αφορά το συνάδελφο Κόρμπι Μίκε, Είχα την τυχαία να προεδρεύω σε εκείνη τη συνεδρίαση. Ήταν κάτι πραγματικά πολύ άσχημο. Έλαβε ποινή από το Προεδρείο, αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όχι εξής του περιεχομένου, αλλά επειδή στη μερίσια διάταξη γράφεται ότι οι ποινές Ε, δεν θα υφίστανται όταν κάτι δεν επαναλαμβάνεται και όταν υπάρχει και αναστάτωση μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Προσπάθησα να αποτρέψω μια τέτοια αναστάτωση. Ωστόσο, καταφέραμε μεταξύ να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι αποδεκτό. εξαιτία τη διαδικασία το να μην ισχύει ε, η περίπτωση ποινή, το θεωρώ λάθο. Όσον αφορά το ερώτημα για την ε, επαγγελματική κατάρτιση. Έχουμε μαθήματα. Η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού θα έχει μαθήματα για άτομα που ασχολούνται με την επιλογή προσωπικού Επίσης, θα γίνουν, ε, θα ληφθούν μέτρα για την σωστή αξιολόγηση των επιδόσεων για να μην υπάρχει αυτός ο ασυνείδητος διαχωρισμός και να μην συνεχιστεί ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό. Θεωρώ ότι και αυτό είναι μια απάντηση σε αυτά που είπατε. Επιπλέον, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει υποχρεωτική εκπαίδευση στο μέλλον για όλα τα μέλη και τους συνεργάτες. Αυτή η ομάδα θα ζητήσει τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμών για θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης στο Ευρωκοινοβούλιο και την ε, δυνατότητα και την αρμοδιότητα της Επιτροπές να μπορούν να εξετάσουν ε, περιπτώσεις καταγγελιών. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. γιατί δεν είναι κάτι αυτονόητο στο Προεδρείο. Η ύπαρξη εμπειρογνωμόνων δεν πετύχαμε αρχικά πλειοψηφία, όμως πιστεύω ότι θα την πετύχουμε. Επίσης, η ενίσχυση της Επιτροπής για την καταπολέμηση των παρενοχλήσεων για την, με την ύπαρξη μιας ενίας επιτροπής που θα το ελέγχει το θέμα αυτό. Αυτό θα ήταν πιο αποτελεσματικό και είναι ένα από τα μέτρα για τα οποία δεν έχουμε ακόμα την πλειοψηφία, που θα πρέπει να επιμείνουμε όχι μόνο για την γενική διοίκηση, αλλά και για τις πολιτικές ομάδες, ώστε όλο το προσωπικό να λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση. Να μην υπάρξουν κενά. Θα ήταν επιθυμητό να υπάρξουν πιο στεναρές ισχυρέ αποφάσεις μέσα σε εκθέσεις, υποχρέωση για όλους τους υπαλλήλους, όλους τους συνεργάτες σε υψηλές θέσεις. Ακόμα δεν το καταφέραμε, αλλά στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία θα το προωθήσουμε και ελπίζω ότι θα το πετύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ Κύριε Αντιπρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία που είχαμε. Πραγματικά κάναμε μια προσπάθεια κατά τη διάρκεια της θητείας μας έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται καλύτερη εφαρμογή τη ισότητα των δύο φύλων. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και στην επόμενη θητεία. Ε, Σημείο 9 της σημερινής διάταξης η μελέτη για το gender mainstreaming ε, στις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε τώρα μια παρουσίαση της μελέτης για το θέμα αυτό. Επίσης ε, έχουμε εδώ αυτούς που εκπώνησαν τη μελέτη αυτή σήμερα. Πρώτα απ' όλα θα δώσω το λόγο στο συντάκτη της παρουσίασης αυτής, τη Μανουέλα Σάμεκ Λοντοβίτσι. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα σας παρουσιάσω μια επικαιροποιημένη εκδοχή μιας προηγούμενης μελέτης που έλαβε χώρα το 2014 σε ό,τι το σε ποιο βαθμό η Επιτροπή ΦΕΜ και τα άλλα όργανα που ασχολούνται με το gender mainstreaming στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζουν αυτές ε, τις ε, πρακτικές ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μιλάμε για την περίοδο Ιούλιο 2017 με Ιούλιο 2018. Έχουμε λοιπόν εδώ μια σφαιρική εικόνα του πώς το gender mainstreaming εφαρμόστηκε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξετάσαμε ιδιαίτερα της ε, δραστηριότητε της Επιτροπής ΦΕΜ, Επιτροπής Γυναικών, καθώς ε, και το δίκτυο ε, για το gender mainstreaming και, η ομάδα και την ομάδα ψηλού επίπεδου. Εξετάσαμε επίσης ποιες είναι οι νομοθετικές και μη νομοθετικές δραστηριότητες της Επιτροπής ΦΕΜ, καθώς και εξετάσαμε για την εξέλιξη της παρουσίας των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό το τελευταίο σημείο παρουσία των γυναικών. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 2018 περίπου κάτι παραπάνω από το 1 τρίτο του συνόλου των μελών. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο, ε, το προηγούμενο κοινοβούλιο, πολύ μικρή αύξηση, 0,3%. Όμως υπάρχει μια μεγαλύτερη αύξηση σε ό,τι αφορά την παρουσία των γυναικών σε θέσεις ε, λήψη αποφάσεων. Πέντε γυναίκες αντιπρόεδροι από τους 14, ενώ ήταν μόλις τρεις στην 7η ε, θητεία και οι μισές επιτροπές, ε, τις μισές επιτροπές προεδρεύουν γυναίκες. Είναι και αυτό μια βελτίωση, παρότι εξακολουθούν να υπερπροσωπούνται οι γυναίκες στις υψηλόβαθμες θέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, η σύνθεση των φύλων στις διάφορες επιτροπές ε, ε, ποικίλει, ανάλογα με την επιτροπή. Κάποιες επιτροπές ε, ε, είναι λιγότερο από 20% οι γυναίκες, όπως η ΚΟΝΤ και η ΑΦΕΤ, και μόλις σε τρεις επιτροπές το ποσοστό αυτό ξεπερνάει το 50%. ΦΕΜ, ΠΕΤΗ και Λίμπε Εξακολουθούν να εκπροσωπώνται πολύ ισχνά σε θέσεις διαχείρισης του Κοινοβουλίου γυναίκες. Μόλις δύο από τις 12 ε, αναπληρωτές, γενικοί διευθυντές, 2 στις 12, λιγότερο δηλαδή από 17%, όταν ο δικός χάρτης ε, της ομάδας του επίπεδου προέβλεπε έναν στόχο της τάξης ε, του 30% για το 2019, στα μισά είμαστε εμείς και οι μισοί από τους γενικούς διευθυντές, ε, οι μισές από τους γενικές διευθυντές αποτελούνται μόνο από άντρες και μόλι σε τέσσερι υπάρχουν περισσότερε γυναίκε από άντρε. Βλέπετε λοιπόν εδώ την υποεκπροσώπηση. Επίση οι γυναίκε υποεκπροσωπώνται μεταξύ των ομιλητών στι ακροάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζουμε λοιπόν στην επόμενη θητεία να υπάρξει βελτίωση, αν και δεν είμαι και τόσο βέβαιη. Λοιπόν, η εξέλιξη του gender mainstreaming στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση βλέπουμε ότι υπάρχει μια βελτίωση παρότι αυτή η βελτίωση είναι αργή. Υπάρχει ένα νομικό, θεσμικό πλαίσιο που υποστηρίζει το gender mainstreaming πέρα από την Επιτροπή Γυναικών που έχει και τον κεντρικό ρόλο σε νομοθετικό και μη νομοθετικό επίπεδο. Υπάρχει το δίκτυο για το gender mainstreaming, πολύ σημαντικό, μιας και υποστηρίζει την εφαρμογή του gender mainstreaming στις άλλες επιτροπές έχετε δηλαδή να συμπληρώσει αποτελεσματικά το ρόλο της ΦΕΜ και βεβαίως η ομάδα υψηλού επίπεδου ε, για την ισότητα των δύο φύλων και την ποικιλομορφία που προωθεί το gender mainstream βεβαίως στα πλαίσια των δομών και των οργάνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προετοίμασε τον οδικό χάρτη για να αυξηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών στις ε, μεσές και υψηλόβαθμες θέσεις διαχείρισης 40% στο 2020. Αυτός είναι ο στόχος, δεν ξέρω αν θα επιτευχθεί. Υπάρχει και ένα υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής, ε, των, ε, μάλλον συμπερίληψης των προτάσεων της Επιτροπής Γυναικών και των τροπολογιών της σε άλλες εκθέσεις άλλων επιτροπών. Όμως βεβαίως πολλά μένουν να γίνουν υπάρχει σίγουρα περιθώριο βελτίωση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το συντονισμό μεταξύ των διαφόρων οργάνων που υποστηρίζουν και προωθούν το gender mainstreaming στο κοινοβούλιο. Τώρα, σε αυτό το πίνακα δεν ξέρω αν το βλέπετε, συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση ούτω ή άλλω, έχετε ένα κατάλογο με τα βασικά θεσμικά βήματα που έγιναν στο Κοινοβούλιο από το 2003 και μετά για το gender mainstreaming. Και βλέπετε τα τελευταία χρόνια από το 2016 και μετά δηλαδή, έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Ψήφισμα για το gender mainstreaming, ορισμός ενός ε, μόνιμου εισηγητή, ε, κριτές γραμμές ε, για μια γλώσσα που να είναι ουδέτερη σε ό,τι αφορά το φύλλο, ε, παρουσίαση για τις ό,τι των δύο φύλλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, στη Γραμματεία πιο συγκεκριμένα και βεβαίως το ψήσιμο του της Ολομέλειας για το Gender Mainstreaming που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο φέτος. Πολλά λοιπόν έχουν γίνει. Σε θεσμικό επίπεδο. Τώρα, τι έχει κάνει η Επιτροπή Γυναικών, η Επιτροπή ΦΕΜ για αυτό το έτος, έτσι πάντα. Ε, εάν το συγκρίνουμε με την περίοδο του 2014, την περίοδο του 2011-2013, εν πάση περιπτώσει, ε, έχουμε περισσότερα, μεγαλύτερη έγκριση ε, τροπολογιών και προτάσεων τη επιτροπή ΦΕΜ σε άλλε επιτροπές, όμως σε αυτή την περίοδο η Επιτροπή ΦΕΜ δεν ε, εκπώνησε κάποιο νομοθέτημα. Σε αυτή την περίοδο η Επιτροπή ΦΕΜ έχει ε, ε, προετοιμάσει εννέα εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας, ε, ολική παρενόχληση, βία κατά των γυναικών, αλλά και κάποια ζητήματα τα οποία δεν σχετίζονται συνήθω με, με την ισότητα των δύο φύλων, κλιματική αλλαγή, παραδείγματο χάρη, ο τομέα των μέσων ενημέρωση. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει παρέμβαση πλέον και σε άλλου τομεί πολιτική και αυτό είναι σημαντικό. Διότι όταν μιλάμε για gender mainstreaming, το mainstreaming σημαίνει ότι πρέπει το θέμα των δύο φίλων να τη χάνει προσοχής ε, και σε άλλους ε, τομείς, όχι μόνο σε εκείνους τους προφανείς. Ε, υπήρξε και μία, μία, μία μη νομοθετική έκθεση για τη σύμβαση της Ινσταμπούλ ε, για την πρόληψη και την σύγκριση της βίας κατά των γυναικών, 13 νομοδοτήσεις με 259 προτάσεις κυρίως βέβαια στους συνηθισμένους ε, τομείς που σχετίζονται με την ισότητα των δύο φύλων ε, και επίσης 13 ε, τροπολογίες σε 6 διαφορετικές εκθέσεις. Βλέπουμε εδώ τώρα σε ποιο βαθμό αυτές οι προτάσεις στις νομοδοτήσεις και οι τροπολογίες έχουν εγκριθεί από τις άλλες επιτροπές. 13 εκθέσεις ε, ε, και πάνω από 200, 259 συνολικά προτάσεις έχουν υποβληθεί σε 7 επιτροπές και όπως βλέπετε 47,5% αυτών των γνωμοδοτήσεων ε, έγιναν αποδεκτές, αυτό, των τροπολογίων ε, των προτάσεων έγιναν αποδεκτές είτε εν μέρη είτε ε, πλήρως. Βλέπετε εδώ τον αριθμό των προτάσεων που έγιναν αποδεκτές. Εδώ βέβαια υπάρχει απόκληση από επιτροπή στην επιτροπή. Το πιο ψηλό ποσοστό ε, αφορά την επιτροπή Γιούρι και το χαμηλότερο αφορά την Επιτροπή Προπολογισμού και είναι αρκετά χαμηλό επίσης το ποσοστό ε, έγκρισης στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δούμε γιατί ε, συμβαίνει αυτό. Το άλλο ζήτημα είναι οι τροπολογίες gender mainstreaming που είναι πολύ εστιασμένες, πολύ συγκεκριμένες ε, για πολύ συγκεκριμένα θέματα, αυτές έχουν υψηλότερο ποσοστό έγκρισης, 63% έγιναν αποδεκτές εν μέρη ή εν όλο, σε πέντε διαφορετικές επιτροπές όπου υπευλήθησαν και πάλι το πιο, χαμηλό, το, το πιο χαμηλό ποσοστό αφορά την Επιτροπή ΕΚΟΝ, όλα τα θέματα που έχουν κάνει τον τα οικονομικά ζητήματα, ε, όλα αυτά εκεί είναι δύσκολο ε, να επιβάλλει κάποια προσέγγιση gender mainstream. Χαμηλό το ποσοστό και ε, στην, στην απασχόληση, στην ΕΜΒ μάλλον, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, μόλις 15%. Το υψηλότερο ποσοστό πάντως αφορά την Επιτροπή Απασχόλησης είναι πιο εύκολο εκεί βέβαια. και καταλαβαίνει καλύτερα ο κόσμος γιατί το θέμα της όντως των δύο φύλων είναι κρίσιμο. Το ίδιο και στην Επιτροπή Ελευθερίας, Ελευθεριών και στην Επιτροπή Αναφορών. Ε, θέλησαμε να δούμε αν υπάρχει ένα συσχετισμό μεταξύ του ποσοστού αποδοχής αυτών των προτάσεων και των τροπολογιών της Επιτροπής ΦΕΜ. Εάν λοιπόν αυτό συνδέεται με την παρουσία γυναικών ε, σε αυτές τις επιτροπές. Αν δηλαδή οι επιτροπές με μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών αποδέχονται πιο εύκολα ε, προτάσεις από την Επιτροπή ΦΕΜ. Δεν προκύπτει όμως κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σχέση. Από ό,τι φαίνεται είναι πολύ πιο σημαντικό ε, το ποιος είναι ο εισηγητής και όχι τόσο η παρουσία γυναικών. Ένα άλλο που εξετάσαμε είναι το θέμα των πολιτικών ομάδων. Κατά πόσο δηλαδή ε, ο συγητή ΦΕΜ ε, είναι ο ίδιο στην την πολιτική ομάδα με αυτόν τη άλλη επιτροπή. Ούτε εκεί όμω προκύπτει κάτι τέτοιο. Ε, το τελικά το καθοριστικός ρόλος είναι πόσο σημαντικό είναι το θέμα, πόσο αφορά το gender mainstream. Δηλαδή για τα ζητήματα εκείνα που θεωρούνται ότι σχετίζονται με το θέμα, τα θέματα των δύο φύλων, εκεί οι τροπολογίες περνάνε. Ε, σε άλλους τομείς, σε άλλα πεδία, είναι πολύ δύσκολο. Να γίνουν αποδεκτές, διότι δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση για το πόσο σημαντικά είναι αυτά τα θέματα και πώς το θέμα της όντας των δύο φύλων και η σχετική προσέγγιση θα μπορούσε να βελτιώσει τελικά την ε, πολιτική. Συστάσεις τώρα. Οι συστάσεις είναι παρενθερείς με αυτές που είχαμε προβλέψει πριν από τέσσερα χρόνια. Εξετάζοντας το τελευταίο ψήφισμα, αυτό που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο φέτος, αυτό επιβεβαιώνεται. Το ψήφισμα προσπαθεί να υποστηρίξει εδώ ένα πιο ισχυρό ρόλο για την Επιτροπή Γυναικών. Ένα θέμα λοιπόν είναι το θέμα του καθεστώτος τη Επιτροπή ΦΕΜ. μια οριζόντια επιτροπή έχει δηλαδή μια ευρεία δυνατότητα παρέμβασης σε όλους τους τομείς πολιτικής, αλλά σπάνια ε, είναι η ίδια η Επιτροπή ΦΕΜ επικεφαλής στην νομοθετική διαδικασία. Είναι μεταξύ των ε, άλλων επιτροπών ε, σε μια υβριδική κατάσταση Δηλαδή μπορεί κάποιο να επηρεάσει, μπορεί να επηρεάσει αυτή η επιτροπή τι αποφάσει που παίρνουν από άλλε επιτροπέ, αλλά δεν παίρνει η ίδια τι αποφάσει. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο επιτυχεί ε, στο να έτσι ώστε η Επιτροπή Γυναικών να επηρεάσει περισσότερο. Ε, να πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλο τη Επιτροπή ΦΕΜ και στη σύσταση άλλωστε αναφέρεται ότι οι άλλε επιτροπέ θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τις προτάσεις και τις ε, τροπολογίες της Επιτροπής ΦΕΜ. Είναι σημαντικό οι συγητές ΦΕΜ έτσι να είναι ισχυροί, να, είναι, να μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και βεβαίως ε, το θέμα της όρτης των δύο φύλων και το πόσο αυτό το θέμα ε, επικρατεί στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική ατζέντα. Για να μπορέσει λοιπόν να βελτιωθεί όντως αυτή η προοπτική ισότητα των δύο φύλων σε τομεί πολιτική που δεν θεωρούνται συνήθω ε, σχετικοί, ε, είναι σημαντικό η Επιτροπή ΦΕΜ να συνεχίσει ε, να ε, προωθεί τη συζήτηση αυτή. Πώς δηλαδή όντω η προοπτική της ισότητα των δύο φύλων μπορεί όντω να βελτιώσει την λήψη αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο, ιδιαίτερα στου τομεί εκείνου που δεν θεωρούνται σχετικοί με τις ισότητα των δύο φύλων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα προεκλογικό προγραμματισμό με εκθέσει πρωτοβουλία και εισηγητέ που θα εμπλέκουν και άλλε επιτροπέ στο μέτρο του δυνατού σε κοινέ ε, εκθέσει. Είναι πιο εύκολο έτσι να προωθήσουμε αυτή τη νέα προσέγγιση και γενικά να ε, προωθήσουμε την, ευρεία, την ευρύτερη συζήτηση, τη δημόσια συζήτηση, όχι μόνο στο Κοινοβούλιο, εκτό Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα στου τομεί εκείνου όπω ήταν των δύο φίλων δεν θεωρείται σχετική επαναλαμβάνω, πρέπει να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση. Πολύ, η ευαισθητοποίηση. Πολύ σημαντικό αυτό, όχι μόνο για τις γυναίκες, για όλους. Για να βελτιωθεί ο ρόλος της ΦΕΜ, βεβαίως υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος της στην νομοθετική, στις νομοθετικές προτάσεις και εδώ παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο βεβαίως ε, ο ρόλος της Προέδρου και της Γραμματείας ε, θα πρέπει να υπάρξει ένα στρατηγικό σχεδιασμός ε, συνεργασία με, άλλους, με άλλε επιτροπές ε, για εκθέσει πρωτοβουλία της ΦΕΜ για να υπάρχει ένας μηχανισμός προδέσμευσης, αν θέλετε, για να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και μεγαλύτερη προσοχή σε ζητήματα των δύο φύλων. Υπάρχει ανάγκη καλύτερης επιλογής ε, των γνωμοδοτήσεων, διότι η Επιτροπή ΦΕΜ, αυτό το είδαμε και στην προηγούμενη έκθεση, οι άνθρωποι εκεί έχουν πολλή δουλειά, διότι πρέπει να παρέμβουν για τα πάντα και ορισμένε φορέ δεν προλαβαίνουν. Συνήθω είναι και μέλη άλλων επιτροπών. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια επιλογή, επιλογή για να εστιάσει σε, στα, στις προτεραιότητες της Επιτροπή ΦΕΜ και θα πρέπει να υπάρξει και συμμετοχή των μελών του Κοινοβουλίου που δεν είναι μέλη της Επιτροπής ΦΕΜ στις τροπολογίες αυτές για το gender mainstreaming να αυξηθεί και με αυτόν τον τρόπο ευαισθητοποίηση. Υπάρχει και μία ανάγκη, αναφέρεται αυτό στο τελευταίο ψήφισμα, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί δηλαδή, η ανάγκη καλύτερου συντονισμού μεταξύ των τριών οργάνων, δηλαδή το δίκτυο, η ομάδα του επίπεδου και η Επιτροπή ΦΕΜ. και να ενισχυθεί και ο ρόλος ε, του δικτύου gender mainstreaming διότι αυτή συμμετέχουν και σε άλλε επιτροπέ και μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν την Επιτροπή ΦΕΜ έτσι ώστε να προωθηθούν και να εγκριθούν τελικά οι τροπολογίε του, οι προτάσει του. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι κοινοί στόχοι στου οποίου θα πρέπει να εστιάσουμε και υπάρχει αυτή και η ιδέα τη παρακολούθηση τη εφαρμογή του Χάρτη από την ομάδα υψηλού επίπεδου. Τελειώνοντας, Αυτό το συζητήσαμε και νωρίτερα για τη σεξουαλική υπερενόχληση, Ε, υπάρχει η ανάγκη να ενισχύσουμε τη δυνατότητα εφαρμογής του gender mainstreaming στις επιτροπές, ε, στα όργανα του Κοινοβουλίου, χρησιμοποιώντας εσωτερική και εξωτερική πραγματοδομοσύνη, χρησιμοποιώντας την κατάρτιση και για τα μέλη του Κοινοβουλίου και για το προσωπικό και για τη γραμματεία, να προωθήσουμε νέα εργαλεία όπως αξιολογήσεις αντικτύπου ε, στα, στο θέμα των δύο φύλων ε, και άλλα τέτοια εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί. Να προωθήσουμε λοιπόν τη χρήση των νέων εργαλείων, να προωθήσουμε μελέτες, ε, κατάρτιση και για τη γραμματεία. Αυτά. Ευχαριστώ. Thank you very much. ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος, για την έρευνά σας, για την ε, μελέτη σας. Ευχαριστούμε που την ε, παρουσιάσατε. Δεν ξέρω αν θέλει η κυρία Λόι να πει κάτι. Α, η κυρία Νόιχελ, θέλετε να πείτε κάτι εσείς. Για μία ακόμα φορά σας ευχαριστώ πολύ. Η μελέτη σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική κιόλα. Ε, δίνει μία έποψη γενικά της εργασίας ε, στο Κοινοβούλιο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε την έμφυλη διάσταση. Είναι σημαντικό ε, να μας ακούσουν βέβαια και οι ε, Υπουργοί Οικονομικών, ε, γιατί εγώ έχω δουλέψει στο Υπουργείο Οικονομικών της Λιθουανίας και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι εκεί δεν γίνεται και πολύ μεγάλος λόγος ε, για τις γυναίκες και τις ανάγκες των γυναικών. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε στο νέο κοινοβούλιο ισχυρή παρουσία των γυναικών και θέλουμε και μια επιτροπή φάμε στο επόμενο κοινοβούλιο που θα ε, συνεχίσει τον αγώνα για όλα αυτά τα θέματα. Αυτό ήταν το τελευταίο θέμα στη Μερίσια Διάταξη. Σας ευχαριστώ όλους ε, που συμμετείχατε. Ευχαριστώ ε, Μαρία ειδικά που ήσουν πάντα τόσο στόχο Ευχαριστώ τα μέλη της Γραμματείας. Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι μας παρακολουθούν, μας παρακολούθησαν με μεγάλη προσοχή. Ε, και ευχαριστώ πολύ και την ομάδα της ε, Μαρίας Νόιχερ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους ε, για την σοβαρή δουλειά και είμαι σίγουρη ότι θα ξανασυναντηθούμε τον Ιούλιο σε μια νέα συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ.